Hello everybody. Um, bienvenue. Σας καλωσορίζω λοιπόν. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Θα μιλήσω στα αγγλικά όμως, αν και έχουμε πολλούς Γάλλους. Επειδή έχουμε λέει πρόεδρος πολλούς Γάλλους θα μιλήσω αγγλικά. Χαίρομαι που σας συναντώ όλους εδώ σήμερα Έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες παρουσίες, δικηγόρους, δημοσιογράφους. Today on the topic of Για τον ρόλο των γυναικών στον εκδημοκρατισμό στις κοινωνίες της Μέσης Ανατολής. Ήταν έκπληξη για πολλούς από μας αυτό το οποίο συνέβη στην περιοχή και ήταν επίσης σημαντική έκπληξη το ότι οι γυναίκες πήραν τόσο σημαντικό ρόλο και ήταν πρωτοπόρες οι γυναίκες στις επαναστάσεις αυτές. Ήταν λοιπόν κάτι το πάρα πολύ θετικό. Εξακολουθώ να θαυμάζω και να εκφράζω ακριβώς ε, το σεβασμό μου για τη δύναμη, την εξυπνάδα, την οξύνια την οποία επέδειξαν οι γυναίκες στις περιοχές αυτές τους τελευταίους μήνες και τις τελευταίες δεκαετίες. Αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε είναι να δώσουμε μεγαλύτερη δημοσιότητα σε αυτές τις πρωταγωνίστριες και έτσι οι φωνές των γυναικών να συνεχίσουν να ακούγονται και να μην αχαθούν τις επόμενες εβδομάδες τις προσπάθειες που συνεχίζονται για την αποκατάσταση της δημοκρατίας σε ορισμένες χώρες και στις επαναστατικές διαδικασίες από την άλλη. Δύο ομιλίες καταρχάς από δύο ομιλήτριες και μετά ένα πρώτο πάνελ συζητήσεων. Έχετε μπροστά σας τη σωστή ημερήσια διάταξη. ξέχασα να παρουσιαστώ. Λέγομαι Φραντσίσκα Μπράντνα, είμαι μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών. Είμαι αναπληρώτρια της Επιτροπής Γυναικών και είναι τιμή μου που προεδρεύω στον πρώτο γύρο αυτής της συνάντησης. Θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Καντέρ, καθηγητή στο Καθολικό Πανεπιστήμιο της Λουβά και ε, διευθυντής του ΦΕΡΜΑΚ, του Κέντρου Σύγχρονων Αραβικών Μελετών. Ήταν ε, μέλος της ομάδας εμπειρογνωμόνων για την ΚΕΠΑ και για τον, ε, την ομάδα για την πολιτιστική συνεργασία στη Μεσογειακή περιοχή, Μεσογειακή Λεκάνη. Θεωρείται ένας από τους καλύτερους αναλυτές των σχέσεων ανάμεσα στον Ευρωπαϊκό και τον Αραβικό κόσμο. Χαίρομαι για την παρουσία σας, κύριε Καμέλ. και ευχαριστώ γιατί με την ομιλία σας θα τοποθετήσετε και το πλαίσιο των συζητήσεων που θα ακολουθήσουν. Υπάρχει διερμηνία. Αν δεν μιλάτε γαλλικά, φορέστε τα ακουστικά σας, λέει η Πρόεδρος. Έχουμε σε διάφορες γλώσσες. Δεν πειράζει. Αγαπητοί φίλοι, ευχαριστώ γιατί μου δίνετε την ευκαιρία να αναφερθώ σε κάτι το εξαιρετικό, κάτι το έκτακτο, ένα θέαμα θαυμάσιο το οποίο μας εξέπληξε. Τώρα να μιλήσω γι' αυτό σε 10 λεπτά είναι λίγο δύσκολο. Θα κάνω ό,τι μπορώ όμως για να σεβαστώ το χρόνο τον οποίο μου δώσατε. Ακόμα και οι ικανότεροι των σχολιαστών δεν είχαν μαντέψει ε, το ξαφνικό των εξελίξεων και των επιτευγμάτων των τελευταίων μηνών. Ελπίδες είχαμε. Εγώ στο τελευταίο βιβλίο μου, ο Αραβικός κόσμος, πώς τον εξηγούμε στην Ευρώπη, είχα μιλήσει για την ιδέα της δικτατορίας και για την ιδέα της άνοιξης, της πολιτικής και της δημοκρατίας. Ε, είχαμε όλοι ευχηθεί την αλλαγή. Δεν πιστεύουμε ότι θα υπάρξει αλλαγή το 2011. Αυτά τα οποία συνέβησαν θα γίνουν αντικείμενο στα πανεπιστήμια κοινωνιολογίας, πολιτικής επιστήμης, σαν ένα μείζον συμβάν, σαν μια ιστορική στιγμή στην ιστορία της Νότιας Μεσογείου και του αραβικού κόσμου. Γιατί αυτό και γιατί τώρα Υπάρχουν πολλοί παράγοντες οι οποίοι συμπίπτουν θα έλεγα στην ε, εξέλιξη αυτή. Δεν θα σταθώ στην αυτοπιπόληση ενός νέου 18χρονου Τινησίου που ήταν η στιγμή εκκίνησης αυτής της διαδικασίας θα αναφερθώ πιο πολύ στους διαφορετικούς παράγοντες, δημογραφικές αλλαγές, πολιτιστικές αλλαγές, ε, τεχνολογικές αλλαγές ο αραβικός κόσμος ε, έχει διπλασιάσει τον πληθυσμό του. Έχουμε φτάσει το 2011 σε 330 εκατομμύρια Άραβες. Οι Άραβες κάτω των 21 ετών αντιπροσωπεύουν το 50% του συνολικού πληθυσμού, το, ε, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το 28%. Ο πληθυσμός αραβικός είναι νέος ε, ηλικιακά που σπουδάζει, εκατομμύρια νέων Αράβων σπουδάζουν στα πανεπιστήμια, η παιδεία προχωρά. και οι γυναίκες στις ιατρικές σχολές αντιπροσωπεύουν 56 και 50% του συνόλου των φοιτητών στην Τινησία και στην Αίγυπτο. Αυτοί οι νέοι βέβαια Άραβες διοικούνται από κάποιους προσκολλημένους παλαιού τύπου πολιτικούς ηγέτες. Ο Μουμπάρακ ήταν στην εξουσία από το 81, ο Μπεναλή ήταν 23 χρόνια, ο Καντάφη από το 79 ε, και παρόλα αυτά ο πληθυσμός τους είναι ένας νέος πληθυσμός του οποίου ηγούνται όμως γυρασμένοι και διεφθαρμένοι ηγέτες οι οποίοι ε, λειτουργούν με προπαγανδιστικό, κατασταλτικό και καταπιεστικό τρόπο. Έχουμε λοιπόν και τον πολιτιστικό παράγοντα. Οι Άραβες αυτοί συνδέονται πλέον με τον εξωτερικό κόσμο, γνωρίζουν τι συμβαίνει στον υπόλοιπο κόσμο οι Άραβες. Οι Άραβες λοιπόν επαναλαμβάνω συνδέονται και με τις νέες τεχνολογίες, με τον εξωτερικό κόσμο μέσω του Twitter, του Facebook, του διαδικτύου γενικότερα. Είναι Άραβες οι οποίοι επίσης βλέπουν και ε, πολλές εκπομπές, ε, δορυφορικά κανάλια όπως το Ελαραμπία και ιδιαίτερα το Αλτζαζίρα έπαιξαν σημαντικό ρόλο όχι στην πρόκληση της εξέγερσης αλλά μπόρεσαν να λειτουργήσουν σαν αντικατοπτρισμός των αλλαγών και των εξεγεύσεων. Βλέπουμε λοιπόν και άλλον ένα παράγοντα εδώ, ε, δημογραφικό. Υπάρχουν φυσικά και οικονομικοί παράγοντες. Τα καθεστώτα μετέτρεψαν την οικονομία του μολύβδου σε οικονομία συμμοριακή. Άσκησαν δηλαδή ένα καπιταλισμό συνομωτικό υπέρ του ωφέλους του προέδρου, του αφεντικού, του αρχηγού της κλίκας όπως είδαμε στην Αίγυπτο, στην Τινησία και αυτό οδήγησε σε τρομακτικές α, ε, α, ε, ε, κερδοσκοπικές υπερβολές από τον πατέρα στο γιο με δυναστικό τρόπο, με κληρονομικό τρόπο. Οι χώρες αυτές άλλαξαν, στρεβλώθηκαν, ο πλούτος τους πέρασε από τον πατέρα στο γιο λες και ήταν οικογενειακή υπόθεση και αυτό φυσικά ήταν κάτι το οποίο προκάλεσε εν πολύ στις εξεγεύσεις στον αραβικό κόσμο. Δεν υπάρχει αραβική επανάσταση συνολικά, αλλά υπάρχουν αραβικές εξεγεύσεις. Το πρόβλημα είναι διαρθρωτικό, είναι γυράσκοντα τα καθεστώτα, είναι διεφθαρμένα τα καθεστώτα, είναι δυσλειτουργικά τα καθεστώτα, είναι παρέες και συμμορίες φίλων. πόσο μάλλον που και η βαλβίδα ασφαλείας της μετανάστευσης εδώ και λίγα χρόνια είχε κλείσει γιατί στο παρελθόν επέτρεπε στο να εξάγει κανείς το εξωτερικό το επιπλέον εργατικό δυναμικό. Σε αυτούς τους παράγοντες λοιπόν δημογραφικούς οικονομικούς θα πρέπει να προσθέσουμε και τον κατασταλτικό χαρακτήρα των καθεστώτων με τάσεις διδακτορικές με μείωση των δικτών εκδημοκρατισμού τα τελευταία χρόνια και τον πολλαπλασιασμό κατασταλτικών μέτρων και μέτρων ελέγχου. Αυτοί είναι οι παράγοντες λοιπόν. Τώρα είναι το πώς. Πώς οι νέοι Ε, που προέρχονται από πόλεις, γιατί άνω του 60% προέρχονται από αστικές περιοχές, είναι μορφωμένοι χωρίς ε, ε, καθοδήγηση πολιτική, χωρίς καθοδήγηση κομματική. Οι νέοι αυτοί είχαν εκφραστεί με σύγχρονο τρόπο για την αξιοπρέπεια, για την, για την ελευθερία, χωρίς Ισλαμικά συνθήματα, χωρίς το Κοράνι, αλλά ονειρεύονται οι νέοι του αραβικού κόσμου όπως και οι νέοι της Ευρώπης. Δεν είναι μόνο γανακτισμένοι, αλλά είναι εξεγερμένοι, βλέπουν ότι ο κόσμος τους είναι παγιδευμένος σε αντιδημοκρατικές δομές. Δεν υπήρχε πλαισίωση των νόων αυτών και αυτό φυσικά διευκολύνει την ανάκτηση και την αλωτρίωση των στόχων τους. Οι νέοι αυτοί παρόλα αυτά χρειάστηκε να συνεργαστούν μεταξύ τους και έτσι κατέριψαν τα καθεστώτα ε, του Μπεναλή και του Μουμπάρακ σε συνεργασία με το στρατό. Εκεί που ο στρατός δεν ακολούθησε βλέπουμε ότι οδηγηθήκαμε σε ένα εμφύλιο πόλεμο με ένα καθεστώς το οποίο βομβαρδίζει τον ίδιο του τον πληθυσμό και με τους Λιβύους εξεγερμένους οι οποίοι έχουν γίνει επαναστάτες και αναγκάζονται να χρησιμοποιήσουν τα στρατιωτικά μέσα για να μπορέσουν να πετύχουν τους στόχους τους. Οι εξεγεύσεις οι αραβικές έχουν ειδικά χαρακτηριστικά και αυτό αποδίδεται στα ειδικά χαρακτηριστικά των διαφόρων κρατών. Εκεί όπου τα κράτη είχαν ουσιαστικές κρατικές μηχανές μπόρεσαν να χρησιμοποιήσουν το πετρέλαιο για να τροφοδοτήσουν τη λειτουργία τους. Εκεί όπου τα κράτη είχαν ένα στρατό πιστό μπόρεσαν να αντισταθούν αλλά αυτό φυσικά θέτει στην επιφάνεια τον κίνδυνο σειράξεων με χιλιάδες θύματα. Εκεί όπου τα καθεστώτα ήταν αστυνομικά όπως στην Αίγυπτο και στην Τινησία τότε είδαμε τι συμβαίνει, ε, βλέπουμε το παράδειγμα της ευτυχούς επανάστασης στην ε, Τινησία και το αντιπαράδειγμα στην περίπτωση της Συρίας. Οι νέοι και οι γυναίκες έπαιξαν σημαντικό ρόλο οι γυναίκες και στην Τίνιδα ήταν πρωταγωνίστριες και στο ε, Κάιρο είδαμε τις γυναίκες στην πλατεία Ταχρήρ έσπασε το μύθο που ε, σοβεί στον δυτικό κόσμο ότι η γυναίκα είναι αποκλεισμένη στο νοικοκυριό της μέσα και δεν ασχολείται με τα κοινά. Ε, δεν έχει πράγματι πολιτικά δικαιώματα αλλά κατέκτησαν οι γυναίκες των αραβικών χωρών πολλές εξουσίες μέσω της παιδείας τους, μέσω της δράσης τους στον τομέα της αγοράς της εργασίας, μέσω της δημογραφικής αλλαγής τους, ε, μπόρεσαν να αποδείξουν με θάρρος, με αξιοπρέπεια, πόσο οι γυναίκες αυτές ήταν σημαντικοί πρωταγωνιστές της αλλαγής. Το είδαμε στην Τινησία, το είδαμε στην Αίγυπτο, δυστυχώς στη Λιβύη, το βλέπουμε λιγότερο αυτό. αλλά στην Τινησία οι Τινήσιες διαδηλώνουν μαζί με τους άνδρες τους στον ίδιο βαθμό. Τι θα γίνει τώρα στο μέλλον. Αγαπητοί φίλοι, οι άνδρες και οι γυναίκες γράφουν ιστορία, αλλά ταυτόχρονα δεν γνωρίζουν ποια είναι η ιστορία την οποία συγγράφουν. Ο δρόμος του μέλλοντος δεν θα είναι στρωμένος με ροδοπέταλα και η μεταβατική φάση θα είναι πολύ δύσκολη με δύο βασικούς κινδύνους. Ο, ο πρώτος είναι ο στρατός να κατάσχει τις κατακτήσεις και να υπάρξει ανάκτηση των κατακτήσεων αυτών είτε από Ισλαμικές δυνάμεις είτε από εκπροσώπους του παλαιού καθεστώτος. Η στάση των νέων ανδρών και γυναικών εδώ είναι σημαντικό. Διαδήλωσαν για να έχουν μια ζωή με αξιοπρέπεια, με προοπτικές, με δυνατότητες ε, ε, απασχόλησης για να μπορέσουν να ολοκληρωθούν σαν πολίτες. Ένα τέτοιο καθεστώς βέβαια σημερινό επαναστατικό δεν δημιουργεί θέσεις απασχόλησης. Ε, αυτό δείχνουν οι ιστορικές εμπειρίες. Ότι ότι μετά από κάποιες αλλαγές σε τέτοιο μεγάλο βάθος η οικονομία περνάει σε μια κάποια ύφεση που μπορεί να κρατήσει και τρία και τέσσερα και πέντε χρόνια δείχνουν οι εμπειρίες από τη Λατινική Αμερική. Μετά βέβαια και εφόσον η δημοκρατία έχει πλέον κατησχίσει υπάρχει μια οικονομική ανάπτυξη και θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση όχι μόνο οικονομικά να στηρίξει τα κινήματα αυτά αλλά να θεωρήσει τις χώρες αυτές ουσιαστικούς εταίρους και να μην ακολουθήσει μια ευρωπαϊκή πολιτική πατερναλιστική η οποία αρκείται στο να πληρώνει τα καθεστώτα αυτά με χρήματα τα οποία δεν χρησιμοποιούνται πάντα για τον σωστό του στόχο. Λοιπόν, οι γυναίκες υφίστανται πάρα πολλές διακρίσεις ακόμα και σήμερα ε, θα έλεγα ότι οι πρώτες, ε, ε, γυναίκες, οι πρώτες χώρες που υπέγραψαν τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Γυναικών ήταν η Αίγυπτος και η Εμένη πριν 20 χρόνια. Αλλά οι υπόλοιπες χώρες καθυστέρησαν πάρα πολύ. Θα ήθελα τώρα λοιπόν οι αραβικές χώρες σε σχέση με τους άνδρες και τις γυναίκες που επέδειξαν τεράστιο θάρρος να υπογράψουν ε, ε, την σύμβαση έτσι ώστε οι γυναίκες να πάρουν μέρος στην δημιουργία ενός νέου κόσμου και να μην ισχύει αυτό το οποίο πίστευαν στην Δύση ότι ο αραβικός κόσμος δεν αλλάζει. Et vous m'avez déjà euh, fait la liaison pour euh, le prochain... Euh, μου δώσατε το θέμα για την επόμενη παρουσίαση. Παρουσιάζω τον ε, καθηγητή Φλίντεμαν που είναι το μέρο του Σούντα που είναι η Ένωση για την Εξάλληψη κάθε είδους διακρίσεων κατά των γυναικών, ΣΥΝΤΟ. Πάρα πολύ σημαντικό έγγραφο για τα ανθρώπινα δικαιώματα στα Ηνωμένα Έθνη. Ο κύριο Φλίντεμαν, θα μας κάνει μια γενική παρουσίαση όσον αφορά την επικύρωση εφαρμογή ε, των ε, ιδεών του ΣΕΝΤΑΦ στη Βόρεια Αφρική. Έχετε 10 λεπτά στη διάθεση σας, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Είναι σίγουρα μεγάλη τιμή και προνόμιο να συμμετέχω σε αυτό το σεμινάριο και θέλω να αποτίσω φόρο τιμή σε όλες τις γυναίκες και εκείνους που εργάζονται και εργάστηκαν και συνεχίζουν να εργάζονται για την αλλαγή. Στα 10 μου λεπτά στην παρέμβασή μου θα επικεντρωθώ πραγματικά σε κάποια πέντε θέματα. Πρώτα απ' όλα σε σχέση με τη σύμβαση, μετά για την επικύρωση, την συμμετοχή και εμπλοκή μη κυβερνητικών οργανώσεων και σημαντικά για τις διεργασίες με κάποιες, κάποιους προβληματισμούς και σκέψεις για αυτή τη σύμβαση ως εργαλείο μέσο για την αλλαγή. Πρώτα επί της ουσίας της σύμβασης. Η σύμβαση αυτή είναι μοναδική, διότι είναι μια ασυμμετρική ε, σύμβαση καλύπτει όλα τα θέματα σε σχέση με την αρνητική διακριτική μεταχείριση των γυναικών. Δεύτερον, καλύπτει την αρνητική διακριτική μεταχείριση και στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Τρίτον, η σύμβαση αυτή υποχρεώνει τα κράτη-μέλη που είναι συμβαλόμενα μέρη να άρουν κάθε μορφή αρνητικής διακριτικής μεταχείρισης εις βάρος των γυναικών. Δεσμεύει όμως τα κράτη να βελτιώσουν και την κατάσταση των γυναικών. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και μοναδικό το ότι η σύμβαση αυτή υποχρεώνει τα συμβαλόμενα κράτη να αντιμετωπίσουν τα αίτια και να επανορθώσουν τα αίτια της αντικής διακριτικής μεταχείρισης βάρος των γυναικών που τόσο συχνά βασίζονται σε θρησκευτικές ή πολιτισμικές πρακτικές και παραδόσεις. Εποπτεύεται από την Επιτροπή ΣΥΔΟ η σύμβαση αυτή που συναπαρτίζεται από ανεξάρτητα μέλη από όλο τον κόσμο από τα διάφορα συμβαλόμενα μέρη, από τα 186 κράτη που είναι συμβαλόμενα μέρη. Υπάρχουν έτσι διαργασίε που προβλέπονται στην σύμβαση αυτή και έχουμε την αναφορά ανακράτος, State Reporting Procedure. Θα επανέλθω σε ένα λεπτό. Το 1999 η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υιοθέτησε ένα εθελοντικό πρωτόκολλο στη σύμβαση αυτή, όπου η διαδικασία ατομικής αναφοράς και μια διαδικασία διερεύνηση, συμπεριλαμβάνονται. 101 κράτη-μέλη έχουν επικυρώσει το πρωτόκολλο αυτό. Δυστυχώ όμω μόνο δύο από τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, η Τινησία και η Λιβύη. Είναι σημαντικό και αυτό. Και εν τέλει, για αυτό το θέμα, η σύμβαση αυτή έχει την εντολή να συντάξει, να συντάσει και να διατυπώνει σημαντικές συστάσεις. Σημαντικό για την, ε, ε, τον διαφωτισμό των εμπλεκόμενων μερών. Και αναφέρομαι σε ένα, στην Γενική Σύσταση Υπαριθμών 19 που αναφέρεται στο θέμα της βίας κατά των γυναικών. Η βία κατά των γυναικών χαρακτηρίζεται ως μια μορφή αρνητικής διακριτικής μεταχείρισης εις βάρος των γυναικών και γι' αυτό εμπίπτει, εντάσσεται στο πλαίσιο της σύμβασης αυτής και πρέπει τα κράτη να αναφέρουν τι έχουν πράξει ώστε να αρθεί αυτή η βία κατά των γυναικών ως φαινόμενο. Δεύτερον, επιφυλάξεις. Πολλές από τις χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής έχουν επικυρώσει με εν μέρη επιφυλάξεις. Ε, δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Το κοινό στοιχείο σε αυτές τι επιφυλάξει που υποβάλλονται από τις χώρες της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής είναι ότι δέχονται τις υποχρεώσεις ε, ως κράτη υπό τον όρο και προϋπόθεση ότι όταν θα υπάρξει αντιπαράθεση με τον νόμο της Σαρία, τον Ισλαμικό νόμο, τότε οι αρχές του Ισλαμικού νόμου πριτανεύουν. Κατέστησαν σαφές οι αρχές τις επιτροπές της σύμβασης που συμπεριλαμβάνουν και μέλη από τις Ισλαμικές χώρες ότι τέτοιες επιφυλάξεις είναι σύμβατες με τον στόχο και το πλαίσιο της σύμβασης και γι' αυτό καταρχήν είναι απαράδεκτες και δεν επιτρέπονται τέτοιου είδους επιφυλάξεις. Όμως τέτοιου είδους επιφυλάξεις ποτέ δεν παρακόλλησαν ένα επικοδομητικό διάλογο με τις αντιπροσωπείες των κρατών μελών και κατά τον διάλογο αυτό τα συμβαλόμενα μέρη προτράπηκαν και ενθαρρύνθηκαν να αντιμετωπίσουν αυτό το θέμα αυτών των επιφυλάξεων. Κάποια κράτη το έκαναν αυτό, το Μαρόκο ή την Ισία και σε κάποιο βαθμό προσπαθεί να το κάνει και η Συρία και η Αίγυπτος προσπαθεί επίσης οι επιφυλάξει ε, κυρίως συνδέονται με το άρθρο 2 και το άρθρο 16 σε σχέση με την ισότητα ανδρών και γυναικών μέσα στο πλαίσιο του γάμου και τη οικογένεια. Τρίτον, ΜΚΟ, μη κυβερνητικέ οργανώσει, διαδραματίζουν ένα κέριο, σημαντικότατο ρόλο στην εφαρμογή τη συνθήκη, τη σύμβαση αυτή, με την υποβολή εναλλακτικών ε, αναφορών, σκιωδών εισηγήσεων και αναφορών, αλλά και διαδικασιών εποπτεία στο εγχώριο επίπεδο. Με τι συστάσει όσον αφορά την επιτροπή αυτή τη σύμβαση, όταν θα έχουν αυτέ οι συστάσει υιοθετηθεί. Δυστυχώ δεν υιοθετούνται σε όλες τις χώρες ε, της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής. Δεν είναι δυνατόν παντού στις χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο και να εμπλέκονται οι ΜΚΟ, οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Και βλέπουμε εδώ και τον άτυπο ρόλο τη εργασία που έχουν και έτσι δεν παρουσιάζονται και δεν αποκαλύπτονται ονόματα για παράδειγμα ταυτοτήτων των όσων εμπλέκονται στι ΜΚΟ. Ε, τέταρτο, οι εκθέσεις που πρέπει να υποβάλλονται στην Επιτροπή για την εφαρμογή της ε, και υλοποίηση της ε, συνθήκης. Είναι σημαντικό τέτοιου είδους εκθέσεις να υποχρεώνουν τα κράτη-μέλη να πράξουν, να κάνουν μια ευρύτερη επισκόπηση σε σχέση με τις πολιτικές για τα δικαιώματα του ανθρώπου και τα δικαιώματα των γυναικών που έχουν υιοθετηθεί μέσα στα πλαίσια αυτής της χώρας. Να ταυτοποιούνται τα εμπόδια, τα προσκόμματα που υπάρχουν ώστε να καθίσταται σαφές ε, ως επιχείρημα το θέμα της αντιμετώπισης των επιφυλάξεων. Τέτοιες εκθέσεις συζητούνται σε πολύ, σε πολύ εξειδικευμένο επίπεδο και θα ήθελα να τονίσω εδώ ότι τέτοιου είδους συζητήσεις, τέτοιου είδους διάλογοι, δομημένοι διάλογοι είναι ιδιαίτερα σημαντικοί διότι δεν πολιτικοποιούνται από πλευράς φύσης των συζητήσεων, διεξάγονται από επαΐοντες που προέρχονται από διαφορετικές χώρες του κόσμου και βασίζονται στην σύμβαση, στη συνθήκη αυτή που έχει γίνει ευρέως δεκτή. Μετά από μια εξέταση των εκθέσεων ανακράτος, η Επιτροπή υιοθετεί συστάσεις και ε, ανησυχίες ή μελήματα που μπορούν να έχουν πολύ μεγάλη σπουδαιότητα στο πεδίο της εφαρμογής και υλοποίησης της σύμβασης όσον αφορά τα συμβαλόμενα κράτη-μέλη. Και αυτό όσον αφορά επίσης και τη διατύπωση επιφυλάξεων, όπως ανέφερα και πιο πριν. Μαρόκο, την Ισία, Αίγυπτο, Συρία που καταβάλουν προσπάθειες. Και ένα άλλο σημαντικό παράδειγμα είναι το Κουβέιτ σε σχέση με την επιφύλαξη για το άρθρο 7 της ε, συνθήκης για τα δικαιώματα των γυναικών να συμμετάσχουν στην διαδικασία λήψης απόφασης σε δημόσιο επίπεδο, σε πολιτικό επίπεδο. Επιπλέον, τα συμπεράσματα εν κατακλείδη είναι ένα σημαντικό στοιχείο και υπό άλλη πτυχή όσον αφορά την διεργασία που υφίσταται στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών και αυτή είναι ο οικουμενικός μηχανισμός αναθεώρησης ε, που ε, λειτουργεί μέσα στο πλαίσιο του Συμβουλίου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα όπου ισότιμοι από άλλα κράτη-μέλη ε, εξετάζουν τα θέματα από πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών για τις πολιτικές που ακολουθούνται. Οι συστάσεις που διατυπώνονται και υποβάλλονται από πλευρά της Επιτροπής για τα ίσα δικαιώματα γυναικών και ανδρών εντάσσονται στο πλαίσιο των ε, ε, συστάσεων όσον αφορά το ε, Συμβούλιο για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου μέσα στο πλαίσιο της τακτικής, τακτής αναθεώρησης της Επιτροπής και υποβάλλονται και σκέψεις ε, και προτάσεις ε, που έχουν τη σπουδαιότητά τους ε, για τις χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής. Είχα την ευχαρίστηση να είμαι το μόνο μέλος από την πλευρά μας σε αυτή την Επιτροπή. Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών κατέληξα στο να συνειδητοποιήσω πόσο σημαντικό, πόσο σημαντικό είναι το θέμα της σύμβασης αυτής στα χέρια ΜΚΟ, μη κυβερνητικών οργανώσεων στα χέρια εκείνων από τους κυβερνητικούς κύκλους που θέλουν και επιθυμούν να ε, συνεισφέρουν στην πρόθεση αλλαγών υπέρ των γυναικών και την ευδοκίμηση των αρχών της Χάρτας των Ηνωμένων Εθνών υπέρ των γυναικών. Για αυτούς τους λόγους ελπίζω ότι η σύμβαση αυτή θα συνεχίσει να διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο κατά τα επόμενα χρόνια, κατά το μέλλον, όπου θα, υπάρχουν, θα υπάρξουν σημαντικότατες αλλαγές και στη Μέση Ανατολή όχι μόνο σε αυτή τη σφαίρα αλλά και στην οικονομική σφαίρα, στα πολιτισμικά θέματα, στα πολιτικά και κοινωνικά θέματα και έτσι από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει όχι μόνο αυτή η σύμβαση να χρησιμοποιείται ως μέσο, ως εργαλείο, ως βάση για συζητήσεις με χώρες της Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής αλλά επίσης και στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο, να επικυρώσει, να κυρώσει αυτή τη σύμβαση ή να υιοθετήσει μια διακήρυξη μέσω οποία θα τοποθετείται και θα λέγει ότι δεσμεύεται και εμπλέκεται ώστε να υπάρξει μια βάση για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο των σχέσεων με τις χώρες της Βόρειας Αφρικής και τη μέση Ανατολής ώστε να χρησιμοποιείται αυτή η σύμβαση ως μέσο, ω εργαλείο. Ευχαριστώ. Thank so Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πραγματικά μια πηγή έμπνευσης το ΣΥΡΟ για πολλούς. Και πραγματικά είναι πάλι πολύ ενδιαφέρον που είπατε ότι εργάζεται πάνω στις ερμηνείες ε, του κειμένου. Είναι μια πολύ ζωντανή επιτροπή, η επιτροπή αυτή εδώ και έχετε δίκιο, θα πρέπει να είναι πιο καλά γνωστή και να υποστηριχθεί καλύτερα. Σας ευχαριστώ για τις συμβολή σας. Θα παραμείνετε, ελπίζω, εδώ για ερωτήσεις ενδεχομένως μετά. Περνάμε τώρα στις ε, γυναίκες ομιλητρίες από την περιοχή εκεί. Θα σας δώσω το λόγο μία μετά την άλλη για να περιγράψω την κατάσταση όπως τη βλέπετε. Να δούμε ποιος ήταν ο ρόλος των γυναικών, ποια είναι η κατάστασή του σήμερα, να ακούσουμε σε τι προσβλέπετε, ποιες είναι οι προσδοκίες σας, ενδεχομένως και τι φοβόσαστε και τι περιμένετε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τα κράτη-μέλη να κάνουν για να υποστηρίξουν την εργασία σας. Οι περισσότεροι από εμά εδώ, αν όχι όλοι, θαυμάζουμε αυτό που κάνατε, αυτό που πρέπει επίση ακόμα να γίνει. Θα αρχίσω και θα μιλήσω πάλι καλικά εδώ. Θα ήθελα να ευχαριστώ τους διερμηνείς ε, γιατί δεν έχουν τις ομιλίες των ε, ομιλητών, πράγμα που κάνουμε συνήθως. Θα ήθελα να σας ευχαριστώ πάντως για τη δουλειά σας. Και λυπούμε που θα ξαναμιλήσω γαλλικά τώρα. Θα ήθελα να ότι η κυρία Ζουινή, που είναι μέλος της ε, Τινησιακής Ένωση Δημοκρατών Γυναικών, μάλιστα ιδρυτικό μέλος, και που εργάστηκε διαμακρών σε αυτό το κίνημα. Ήταν επίσης ιδρυτικό μέλος της εφημερίδας Νίσα και που επίσης ε, εκπαιδεύει για τα ανθρώπινα δικαιώματα δικαιώματα των ελληνικών στο Πανεπιστήμιο και ξέρω ότι ακριβώς το Σαββατοκύριακο είχατε στην Νίδα ένα μεγάλο κογκρέσο δυστυχώς δεν μπορούσα να συμμετάσχω αλλά υπήρχε ένα θαυμάσιο πρόγραμμα πάρα πολλά καλά πάνελ, πολύ καλές συζητήσει. Θα σας δώσω το λόγο για να μας πείτε πού βρισκόσαστε, τι σκεφτόσαστε, ποια είναι τα πορίσματα από το Κογκρέσο στο πίσω, και να μας δώσετε και κάποια προοπτική, τι πρέπει να γίνει και τι επιθυμείτε να γίνει. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Όπως είπατε, μόλις οργανώσαμε ένα σεμινάριο για τα δικαιώματα των γυναικών και την δημοκρατική μετάβαση, αλλά εγώ δεν μπόρεσα να είμαι εκεί. Υπήρχαν γυναίκες από όλη την περιοχή και άλλες από την Ευρώπη, από τον Καναδά, για τις ανταλλαγές, γιατί αυτές είναι φεμινίστρες που συναντήσαμε και που θα μας βοηθήσουν για να περάσει η εναλλακτική μας έκθεση τελευταία πριν φύγει ο δικτάτορας, η δική μας οργάνωση υπέβαλε μια καλή εναλλακτική έκθεση για την Επιτροπή ΣΕΝΤΟ. Αυτή είναι η τελευταία έκθεση. Και θυμόμαστε ότι εμείς ζητήσαμε την ισότητα μεταξύ των γονέων για τα παιδιά δηλαδή ίσα δικαιώματα του πατέρα και της μητέρας και ο Υπουργός ε, είχε πει ότι ένα πλοίο δεν χρειάζεται δύο κυβερνήτες. Αυτή ήταν η απάντηση του καθεστώτος Μπεναλή. Αλλά θα σας διαβάσω και ένα εγγραφό που σας αποδεικνύει τι μπορούν να καταφέρουν οι γυναίκες της Τινησίας. Εδώ και 50 χρόνια περίπου μαχόμαστε για τη δημοκρατία και την ισότητα των ευκαιρών. Εδώ και 20 χρόνια η, η ένωση μου, η, την Ισιακή Ένωση Δημοκρατών Υγών, ε, αποφάσισε να μαχηθεί με τις γυναίκες για τα δικαιώματά τους και την αξιοπρέπειά τους. Ακούγοντας αυτά που έχουν να πούν, βοηθώντας τες, προσπαθήσαμε να τους βοηθήσουμε να προωθήσουν αυτά τα αιτήματά τους σε τοπικό, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, συνοδεύοντας τις γυναίκες αυτές για να κερδίσουν τα δικαιώματά τους και την αξιοπρέπειά τους, μπορούμε σήμερα να αποδείξουμε μια αντίσταση γυναικεία εξέλιξη των μορφών της μάχης που ξεκίνησε από τις γυναίκες στις διάφορους τομείς και ενεργή συμμετοχή στην ε, ε επαναστατική διαδικασία. Τα δέκα πρώτα χρόνια της δικτατορίας είχαμε σαν στόχο την απαγόρευση οποιασδήποτε φωνής αντίθετης ε, και εκείνων που μάχονται για την πολιτική. Απ' την άλλη μεριά οι γυναίκες ήταν θύματα ειδική ε, βίας. Ξεκινώντας δηλαδή από την ηθική του την πατριαρχική επιτέθηκε το καθεστώς αυτό σε αυτές και οι γυναίκες αυτές δεν μπορούσαν να έχουν καμία συμμετοχή στην πολιτική, συνδικάτα κλπ. Και εκτός από τη συνήθη ε, καταστολή που σε διάφορες μορφές ε, ήταν ε, θύματα ειδικής βίας σεξουαλικής ε, ε, μοντάζ πορνογραφικών βίντεο και ούτω καθεξής. Αυτές οι επιθέσεις φυσικές και ηθικές είχαν σαν στόχο να τις αποτρέψουν από το να δρούν στο δημόσιο χώρο και συνοδεύονται από ε, καμπάνιες στα ΜΜΕ. Κατά διάρκεια πολλών ετών το καθεστώς προσπάθησε να απομονώσει την ελίτ. Παρ' όλα αυτά προσπάθησε να περικόψει τελείω τα δικαιώματα των γυναικών, να καταβολήψει την τροκομοκρατία και την παράνομη μετανάσταση. Το θαύμα της νησίας, βασίστοσε σε ψευδή στοιχεία και ταυτόχρονα βλέπαμε να επιδεινώνονται οι σχέσεις στις ε, δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις και να προωθείται η διαφθορά και ο νεποτισμός. Η δεύτερη δεκαετία χαρακτηρίστηκε από επιθέσεις κατά των οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων. Πρώτα θέματα το οποίο ήταν οι γυναίκες. Οι γυναίκες είχαν τις πιο ε, κακές θέσεις απασχόλησης και τις λιγότερο καλά πληρονόμονες και σε αυτές προτέθηκαν ε, θέσεις απασχόλησης ε, με περιορισμένα ωράριο στο δημόσιο και εκτός από τα χαμηλά εισοδήματα ήταν μέσα στα πλαίσια των επιχειρήσεων αυτών λόγω της συμμετοχή τους στο RCD το κόμμα του Μπεναλή το λέω σε σεξουαλικές επιθέσεις τις οποίες μας παρουσίασαν. Και ακριβώς ε, λόγω των δηλώσεων αυτών γυναικών των μηνών που εργάζονται στην υπηρεσία για τα ορυχεία ξεκίνησε το ΕΤΕΦΤ μια εκστρατεία σχετική στη δεκαετία του 2000. Κατόπιν είδαμε τις εργαζόμενες στα κλωβιδουλικά να κινητοποιούνται για να προασπίσουν τα δικαιώματά τους στην εργασία, κατέχοντας τα εργοστάσια μαζί με τα παιδιά τους, οργανώντας είναι κάνοντας απεργίες και κλπ. κλπ. Πολλές γυναίκες γνωστές που αποδείξαν μεγάλη τόλμη στην αντίσταση αυτή. Οι νέες αυτές μορφές μάχης που ξεκίνησαν από τις εργαζόμενες στον του τομέα κατά τη διάρκεια των ετών 2000-2006 οδήγησαν την κοινωνία να συνειδητοποιήσει τι γίνεται και να κινητοποιηθεί μαζί τους. Και λόγω της ελληνικής με το κίνημα αυτό και επειδή το συνόδευσε η ΑΤΕΦΤΕ που είχε δημιουργήσει ε, μια μονάδα παρακολούθησης των γυναικών που ήταν θύματα οικονομικών, ε, οικονομικής βίας πέτυχε να πάρει το βραβείο του, το ανθρώπινο βραβείο της Γαλλικής Δημοκρατίας του 2008. Στις μάχες αυτές συμμετείχαν τα συνδικάτα, οι διπλωματούχοι από τα πανεπιστήμια, οι φοιτητέ, γυναίκες και άλλοι. Η δέμιση της, υπηρεσία, της ε, οργάνωσής μας στις μάχες αυτές ήταν τόσο σημαντική που μας ε, κόστισε το πάγωμα των επιδοτήσεων για τα κέντρα που είχαμε και ε, την ε, ε, κλίση της Προέδρου μας στην αστυνομία γιατί επέτρεψε σε νέους να κάνουν τις, οργαν... τις συνεδριάσεις τους μέσα στο δικά μας κτίρια. Αυτή η εξέλιξη οδήγησε στο ότι φοιτήτρες, δικηγόροι, δικαστή δημοσιογράφοι νέοι, κανένας δεν ήταν πια προφυλαγμένος από την αστυνομική βία. Αλλά όσο πιο δυνατή γινόταν η, μηχανή της καταστολής, τόσο πιο έντονη ήταν η αντίσταση. Όλα αυτά που γινόντουσαν εις βάρος τους δεν μπορούσε παρά να κινητοποιήσουν ένα ε, λαϊκό κίνημα το οποίο δεν άρχισε να γίνει. Εκεί, από εκεί ξεκίνησαν και τα ε, γεγονότα στα περιοχή των ενεργείων το 2008 που ξεκίνησε από 13 χείρες που έμειναν πάνω στις ράγες των τρένων του ορχείου επί δύο μήνες και που, με τις οποίες μετά συνεργάστηκαν όλοι οι κάτοικοι της περιοχής εκατοντάδες νέων συνδικαλιστές ε, κρατήθηκαν, συνελήφθησαν, ε, καταδικάστηκαν αλλά οι γυναίκες συνεχίσαν την μάχη τους. Οι γυναίκες αυτές έγραψαν ιστορία με την τόλμη τους και την ε, περηφάνειά τους. Και θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η φίλη Ζάκη Αντιφαΐου μετά που πέρασε τρεις μήνες στην φυλακή επειδή ήταν ήταν μέλος σε μια διαδήλωση δεν μπόρεσε να επανέλθει στη θέση της ως δασκάλα παρά μετά που έφυγε ο διδικτάτορας. Αναφερόμενος στο κίνημα αυτό της περιοχής των αρχείων δεν μπορούμε παρά να ε, αποδίσουμε φόρο τιμή σε όλους τους δικηγόρους. Η δίκη όλων των συνδικαλιστών και όλων αυτών των πολιτικά στρατευμένων ε, δεν μπόρεσε να κρατήσει στη ζωή την Νεζιχά Γιωμά, συντονίστρια της Επιτροπής, η οποία μας ε, άφησε δυστυχώς. Υπάρχουν και άλλοι που έχουν γίνει στόχος της πολιτικής αστυνομίας, όπως η Λίνα Μπενεμεχενή, μετά από την αυτοπιβόληση του νέου Μπουαζιζή. Η καταστολή ήταν ιδιαίτερα μισογενική, ιδιαίτερα σεξιστική. Στο Καστρίν σαν παράδειγμα υπήρξε επίθεση εναντίον των γυναικών ακόμα και σε αραβικά λουτρά. Ένα κοριτσάκι ενός έτους έχασε τη ζωή του εκεί. Υπήρχαν επίσης ε, ύβρις οι οποίες είχαν σαν στόχο να ντροπιαστεί ο πληθυσμός του Ταλά Φώναζαν οι αστυνομικοί, δώστε μας τις γυναίκες σας, τις κόρες σας, τις αδελφές σας. Είσαστε όλοι νόθοι των Αλγερινών, γιατί σε αυτή τη συνοριακή περιοχή, στο δυτικό τμήμα της Τινησίας, η οποία είχε φιλοξενήσει παλαιότερα τους, τους μαχητές του κινήματος για την απελευθέρωση της Αλγερίας και κατηγόρησαν τις γυναίκες τους ότι είναι πόρνες και τα λοιπά. Εν πάση περιπτώσει, ε, κάθε φορά που επιτίθενται στις γυναίκες χρησιμοποιούν την ηθικολογία για να αποτρέψουν τη συμμετοχή των γυναικών στις δημόσιες δραστηριότητες. Παρόλα αυτά συνειδητοποιούμε το πρόβλημα. Αντέξαμε στις 29 του μηνός, διαδηλώσαμε ανοίξαμε τα γραφεία της Ένωσής μας, συνδυαστήκαμε με τις ενώσεις των φοιτητών, πολιορκήθηκαν τα γραφεία της οργανωσής μας από την πολιτική αστυνομία, αλλά η συμμετοχή μας στην μεταβατική προσπάθεια έγινε παρά τις δυσκολίες τις οποίες ε, είχαμε να αντιμετωπίσουμε. Στις 29 Ιανουαρίου κάναμε και μια μεγάλη γυναικεία διαδήλωση απαιτώντα να υπάρχει δημοκρατία και ισότητα και σεβασμός των δικαιωμάτων των γυναικών. Όλοι συνειδητοποιούμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, ξέρουμε ότι τα πρώτα θύματα είναι οι γυναίκες και η παραβίαση των δικαιωμάτων τους, εμείς εμένουμε στα δεδομένα μας όμως Θέλουμε να αρθούν οι επιφυλάξεις σε σχέση με την υπογραφή της Διεθνούς Σύμβασης από τη χώρα μας. Υπάρχουν πολλοί δισταγμοί όμως. Η προσωρινή κυβέρνηση έχει επικυρώσει τις περισσότερες διεθνείς συμβάσεις και την συνθήκη της Ρώμης για τον ποινικό τομέα, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές ε, ε, αντιρρήσεις για την άρση των επιφυλάξεων. Πετύχαμε βέβαια την ισότητα ανδρών γυναικών στους εκλογικούς καταλόγους. Εξακολουθούμε να ευαισθητοποιούμε τις πολιτικές οργανώσεις και τα πολιτικά κόμματα να διασφαλίζουν μια σωστή επαρκή συμμετοχή των γυναικών στις επόμενες εκλογές Συνειδητοποιούμε βέβαια ότι εδώ υπάρχει έλλειψη ενθουσιασμού από τα περισσότερα πολιτικά κόμματα. Αν μου θέσετε ερωτήσεις θα είμαι στη διάθεσή σας. Euh, σας ευχαριστώ για την αναδρομή στο παρελθόν την οποία κάνατε για να δείξετε ποιο είναι το πρόβλημα και για την ανάλυση της σημερινής κατάστασης. Θα υπάρξουν αργότερα ερωτήσεις. Θα ήθελα να καλωσορίσω την κυρία Έλντε η οποία είναι μέλος του προσωρινού Συμβουλίου Μετάβασης στην Λιβύη. Η κυρία Ελντεγκάλη έχει κάνει το διδακτορικό της στο Συνταγματικό Δίκαιο στο Πανεπιστήμιο της Ορβόνης και διδάσκει σε πανεπιστήμιο. Χαίρομαι που είστε ανάμεσά σας σήμερα. Με πάρα πολύ ενδιαφέρον θα περιμένουμε να μας παρουσιάσετε την κατάσταση στη Λιβύη και τι κάνετε για την κατάσταση των γυναικών στην Λιβύη γενικότερα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Ένωση για την πρόσκλησή της για να μιλήσει και η γυναίκα της Λιβύης και να σας πει τι έχει κάνει για την επιτυχία της Επανάστασης. Το πρώτο πράγμα το οποίο θα πρέπει να πούμε είναι να προσπαθήσουμε να δούμε τι συνέβαινε πριν από τις 17 Φεβρουαρίου. Για 42 χρόνια η Λιβύη υπέφερε από έλλειψη ε, θεσμών και συνταγματικών ρυθμίσεων ένα κράτος που έζησε κάτω από την κυριαρχία ενός τρόπου ομιλίας και ενός ανθρώπου κάτω από ένα καθεστώς που ποτέ δεν αναγνώρισε τον πληραλισμό. Μια πλήρη απουσία των δημοκρατικών ενιών και ίσως να έχει φτάσει η στιγμή για να σας δείξουμε σήμερα ότι η Λιβύη είναι η μόνη χώρα η οποία έχει ε, νόμο που απαγορεύει ποινικά την δημιουργία πολιτικών κομμάτων και οι γυναίκες φυσικά υποφέρουν από αυτό και γι' αυτό οι γυναίκες της Λιβύης και ο λαός της Λιβύης απέτησαν να υπάρξουν συνταγματικές μεταρρυθμίσεις. Αυτές οι διαδηλώσεις δεν προκάλεσαν την ανταπόκριση της κυβέρνησης και μάλιστα έγινε ένα αντικείμενο καταστολής ε, με όπλα και με, μάλιστα όχι μόνο με πυροβόλα όπλα αλλά και με μη συμβατικά απαγορευμένα όπλα. Και γι' αυτό πλέον περάσαμε στο να απαιτήσουμε να αλλάξει το καθεστώς. Πρόκειται για μια αυθόρματη ε, εξέγερση και κάποια στιγμή άρχισε να επιταχύνεται έτσι ώστε το, το Συμβούλιο μάλλον Μετάβασης να μετατραπεί στο αντιπροσωπευτικό συμβούλιο για τον λαό της Λιβύης ε, ε, στα μάτια του κόσμου. Πρώτον για να απελευθερώσει τη χώρα, δεύτερον για να διατηρήσει την ενότητα της χώρας με την Τρίπολη σαν πρωτεύουσα, να δημιουργήσει ένα δημοκρατικό κράτος και αυτό μας ανάγκασε στο να προχωρήσουμε στη στρατιωτικοποίηση της Επανάστασης που ήταν στην αρχή μια ειρηνική διαδικασία. Άμα δούμε ποιος είναι ο ρόλος των γυναικών λοιπόν σήμερα διαπιστώνουμε ότι η Λίβια γυναίκα όπως και στις υπόλοιπες χώρες παίζει το ρόλο της, βγήκε από το σπίτι, και μάλιστα στην αρχή οι άνδρες ανταποκρίθηκαν λιγότερο. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο κάποιοι παρατηρητές διασφαλίζει τη συμμετοχή των γυναικών στα, δημοκρατικές, στα δημοκρατικά κινήματα στο μέλλον. Οι γυναίκες της Λιβύης φυσικά ήταν από διαφορετικές προελεύσεις και καταβολές, άλλες φορούσαν νικάμπ, άλλες φορούσαν τζίνς όπως και σε χώρες άλλες όπως η Τινησία και η Αίγυπτος. Οι επαναστάσεις αυτές είναι κοινωνικές επαναστάσεις και ο ρόλος της γυναίκας ελπίζω ότι θα βοηθήσει στο να γεννηθεί μια νέα κοινωνία. Οι γυναίκες ε, επίσης βοήθησαν και στην επικοινωνία με τα διαδίκτυα. Είδαμε γυναίκες όλων των ηλικιών να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις, στις ε, διαδηλώσεις στους αγώνες, είδαμε τις γυναίκες της Λιβύης να θυσιάζουν τα παιδιά τους για ένα καλύτερο μέλλον και για την ανεξαρτησία. Είδαμε γυναίκες γιατρούς, γυναίκες νοσοκόμους να κινδυνεύουν για να φροντίσουν τους εκατοντάδες τραυματίες. Είδαμε επίσης γυναίκες να δίνουν μάχη για να προωθηθούν τα κοινωνικά και πολιτικά μας αιτήματα. Είδαμε λοιπόν ποιος είναι ο ρόλος των γυναικών, πολύ σημαντικός στην επιτυχία της εξέγερσης. Οι γυναίκες αυτές οδηγούν σε μια νέα κατάσταση και θα καταπολεμήσουν και θα υπερισχύσουν του δικτάτορα. Η Λίβια γυναίκα είναι παρούσα, ήταν παρούσα και θα είναι παρούσα. Συμμετέχουν οι γυναίκες και στο Μεταβατικό Συμβούλιο και σε επίπεδο τοπικών αρχών και στα πλαίσια της συμμαχίας της 17ης Φεβρουαρίου. Είναι παρούσα, είναι σύμβουλος και παίρνει μέρος και στις διαδηλώσεις από την πρώτη στιγμή. Αναζητεί την ελπίδα. Η γυναίκα της Λιβύης είναι η μητέρα του μάρτυρα, είναι η μητέρα του θύματος, υποφέρει για το τι συμβαίνει συνεισφέρει γενικά στην πολιτική καθημερινότητα αγκυρωμένη στην πραγματικότητα αλλά και ονειρευόμενη την κατασκευή ενός σύγχρονου μέλλοντος για τις γυναίκες, για τις μητέρες, για τις νέες, αν και η εικόνα της εξέγευσης στη Λιβύη δεν δείχνει ποιος είναι ο πραγματικός της ρόλος. Πολλές γυναίκες έχουν πέσει θύματα στις έχουν πάρει μέρος στις συγκρούσεις τις ένοπλες, είναι παρούσες στις εικόνες, στη τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, έχουν προσφέρει πολλά και να μην ξεχνάμε και την ε, γιατρό Άραμά από την πόλη της Τρίπολης η οποία φιλοξένησε τα θύματα στο σπίτι της να τα θεραπεύσει γιατί φοβόντουσαν να πάνε στα νοσοκομεία για να μην πέσουν θύματα απαγωγής ε, του Καντάφη και δολοφονήθηκε στο σπίτι της στα πλαίσια της ενός εγκλήματος πολέμου. Ε, είναι μάρτυρας πλέον αυτή η γιατρός από την Τρίπολη, δολοφονήθηκε γιατί απλά θεράπευε τους τραυματίες και να μιλήσω και για τις γυναίκες της Αζαουία όταν έτρεχε αίμα στην Βεγγάζη οι άνδρες ζήτησαν να υπάρξει ζιχάντα για την εκδίκηση και η πόλη όλοι εξεγέρθηκε για να εκδικηθεί τη σφαγή της ε, Μπενγκάζη και στην ουσία προχώρησαν σε μια Η μια γυναίκα ηλικιωμένη ανέβηκε στην ε, ταράτσα του σπιτιού της και φώναζε «Αλάχου Ακμπαρ» «Μέγας είναι ο Θεός» και ζητώντας από τους άνδρες και τις γυναίκες να πάνε να πολεμήσουν και αφήστε με και μένα να πάρω βόμβες και να πάω να σκοτωθώ μπροστά όμως τον καντάφε. Γι' αυτό επέτρεψε να τονωθεί το ηθικό των ανδρών και να ανακτήσουν α, τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις στις οποίες ήταν οι δυνάμεις του καθεστώτος. Και στην Αλμιζράτα υπάρχουν γυναίκες οι οποίες θυσίασαν τα παιδιά τους να αναφερθώ και στην περίπτωση της Σουτζαμπάλ Γκάμπη, η οποία ήταν θύμα και πολλοί στην οικογένειά τους επίσης έπεσαν θύματα. Μετά από όλα αυτά που σας είπα για το ρόλο της γυναίκας σε αυτή την εξέγερση βλέπουμε ότι η γυναίκα της Λιβύης έχει πια το δικαίωμα να νιώσει την ελευθερία και την πλήρως ελεύθερη άσκηση των πολιτικών της καθηκόντων και υποχρεώσεων. Η δημοκρατία δεν σηκώνει ημίμετρα. Οι δημοκρατικές αξίες ανήκουν σε όλους και τους άνδρες και τις γυναίκες. Βέβαια τα δικαιώματα κατακτώνται, δεν χαρίζονται και η Λίβια γυναίκα κέρδισε τα δικαιώματά της, την ελευθερία της. Um, thank you Σας ευχαριστούμε πολύ η διαφορά στις παρεμβάσεις δείχνει ότι δεν έχουμε μία αλλά πολλές τέτοιες ανατροπές και επαναστάσεις σε εξέλιξη με τελείως διαφορετικές προϋποθέσεις και πλαίσια και οι γυναίκες συνεχίζουν και αγωνίζονται σε ένα συνολικό αγώνα με τον τρόπο τους για την δικαιοσύνη και την ε, δημοκρατία. Θα σας δώσω, θα ανοίξει και ο γύρος ε, παρεμβάσεων και δεξιά στην άκρη είναι η κυρία Γαμίλα Ισμαήλ που είναι πολύ γνωστή ε, εξέχουσα προσωπικότητα από την Αίγυπτο. Το 1986 αποφύτησε από το Πανεπιστήμιο Καΐρου και έχει δίπλωμα ε, διερμηνίας στο, από το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο του Καΐρου όταν την συνάντησα έξεπλάγινε ότι ήταν τόσο εξαιρετικά τα αγγλικά της. Ε, έκανε εξαιρετική δουλειά όσον αφορά τις κοινότητες στο Κάιρο στο παρελθόν και λόγω αυτής της επίδοσης σε αυτό το έργο της προχώρησε σε σχέση με την, το συμβούλιο που την υποστήριζε και τότε ήταν εκείνη η οποία ήταν, ε, ε, που είχε προκαλέσει τον ε, επικεφαλής του κόμματος της εξουσίας, του, του, του κόμματος που βρισκόταν στην εξουσία και έχει καταβάλει προσπάθειες επί πολλά χρόνια και τώρα συμμετέχει στην, στον αγώνα, πρώτα συμμετείχε στον αγώνα για να αποπευθεί ο Μουμπάρακ και τώρα συνεχίζεται ο αγώνας της για μια νέα δημοκρατική Αίγυπτο. Προσβλέπουμε να ακούσουμε την παρέμβασή σας, παρακαλώ. Ε, well, in the beginning Σας ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα στην αρχή της παρέμβασής μου θα ήθελα να ευχαριστήσω την Τινησιανή Επανάσταση και τις γυναίκες από την Τινησία που μας έδωσαν την πρώτη σπίθα αυτής της Επανάστασης από την Τινησία και την μεταλαμπάδευσαν στην Αίγυπτο. Θα ήθελα να πω και να πω στους ε, Λίβιους ότι θα είναι μακρύς ο αγώνας, μακρύς ο δρόμος και δύσκολος και δυσχερής. Όμως στο τέλος θα υπάρξει φως και ελευθερία και αξίζει το αντίτιμο αυτό να πληρωθεί για την ελευθερία έστω και αν είναι πόδινο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη στάση του και την νωρίς και πρώιμη τοποθέτησή του υπέρ υποστηρίζοντας την επανάσταση στην Αίγυπτο. Αντίθετα είδαμε ότι υπήρχαν πολλές δηλώσεις που δεν είχαν ευθεία πορεία και ε, δεν τοποθετούντουσαν με ευθύ τρόπο όσον αφορά τις ΗΠΑ και την κυρία Κλίντον ως Υπουργό Εξωτερικών για την Επανάσταση στην Αίγυπτο. Θα ήθελα να πω ότι η Επανάσταση στην Αίγυπτο είχε τα, τις πρώτες τις ρίζες που έφταναν μέχρι το 2004 εν σπέρματι. Δώσαμε αγώνες και με ήπιο τρόπο αντισταθήκαμε μεταξύ 2004 και 2011. Συνεχιζόταν η ήπια αντίστασή μας και προσπαθήσαμε με κάθε τρόπο να απελευθερώσουμε τη χώρα μας, την, τους Αιγύπτιους και την ίδια την Αίγυπτο από μια φρικτή, φρικαλέα δικτατορία. Αλλά μια και 7.000 χρόνια ολόκληρα οι Αιγύπτιοι ζούσαν και δεν ήταν σε θέση να γνωρίσουν άλλο καθεστώς παρά μόνο αυταρχικά καθεστώτα για τα, στα τελευταία χρόνια πίστεψαν οι Αιγύπτιοι ότι αν και όταν θα υπάρξει επανάσταση θα δημιουργηθεί και θα προκληθεί από τους Ισλαμιστές το αντίθετο όλοι εξεπλάγησαν ακόμα και εκείνοι που με μεγάλες προσπάθειες ε, είχαν αγωνιστεί τα τελευταία δέκα χρόνια όλοι εξεπλάγημεν για το πως οι πολίτες της Αιγύπτου συμμετείχαν και κινητοποιήθηκαν στο τέλος. Θέλω να σας πω ότι οι γυναίκες σε αυτή την επανάσταση, οι γυναίκες οι ίδιες συμμετείχαν, πήραν τον πρωτοπόρο ρόλο, τον ρόλο προπομπών και πρωτοπόρων για πρώτη φορά. Όχι, μια, όχι μόνο σε μια επανάσταση και σε μια ε, προσπάθεια για ανατροπή και για την κοινωνία των πολιτών, αλλά στην κοινωνία συνολικά Θέλω να σας πω ότι η Αιγυπτιακή Επανάσταση είναι μια λαϊκή επανάσταση των πολιτών, χωρίς κάποια ηγεσία, χωρίς στρατευμένη ε, κομματική ομάδα. Για πρώτη φορά οι γυναίκες ήταν στην πρώτη γραμμή ως στρατηγοί και όχι ως στρατιωτάκια, ως φαντάρι ε, που έπαιρναν εντολές από κάποιους. Θέλω να σας πω ότι ήταν μια αστική επανάσταση σε αντίθεση με την επανάσταση στην Τινησία που ξεκίνησε στα χωριά, η επανάσταση στην Αίγυπτο ξεκίνησε σε τρεις μεγάλες πόλεις, το Κάιρο, την Αλεξάνδρεια και το Σουέζ. Και είμαι υπερήφανη γιατί είμαι μία από εκείνες τις γυναίκες που συμμετείχαν και προετοίμασαν αυτή την επανάσταση ενεργά. Θα ήθελα να σας πω ότι οι γυναίκες μέσα σε αυτό το πλαίσιο δεν είναι φεμινίστριες. Κάνω λόγο για τις γυναίκες γενικά στην Αίγυπτο απλές γυναίκες είμαστε και πιστεύω ότι οι φεμινιστές ή φεμινίστριες που έχουν καταβάλει αγώνες και προσπάθειες κατά τα τελευταία 20 χρόνια, τις δύο τελευταίες δεκαετίες στην Αίγυπτο ή στον Αραβικό κόσμο για να απελευθερώσουν τις γυναίκες και να προασπίσουν και προστατεύσουν τα δικαιώματά τους αυτές οι γυναίκες ήταν μεν μέρος, τμήμα αυτού του κινήματος, αυτής της επανάστασης, αλλά δεν ήταν οι μόνες που οδήγησαν και συμμετείχαν σε αυτή την επανάσταση. Οι γυναίκες ξεπέρασαν τα στενά όρια των ιδεών ή των πλαισίων φεμινιστικών αρχών που γυναίκες εργάζονται αποκλειστικά για να προστατέψουν δικαιώματα γυναικών και να αποκτήσουν γυναικεία δικαιώματα. Εμείς συμμετείχαμε και δράσαμε σε αυτή την επανάσταση και δεν ξέρω γιατί όπως, με τους, όπως και οι άντρες. Οι γυναίκες και οι άντρες ως πολίτες που ζητούσαν να υπάρξουν πολιτικές αλλαγές και που θέλανε την επανάσταση αυτή να την προχωρήσουν ένα βήμα παραπέρα, ένα βήμα πιο κάτω, να γίνει μια κοινωνική επανάσταση, μια επανάσταση αρχών, μια επανάσταση αξιών κατά μιας συντηρητικής κοινωνίας. Μια επανάσταση όπου γυναίκες, για τις γυναίκες σήμερα δεν θα ήταν μια επανάσταση για να προστατέψει μόνο δικαιώματα γυναικών και να δημιουργήσει ένα περιθώριο δικαιωμάτων μόνο για τις γυναίκες, αλλά θα ήταν μια απελευθερωτική επανάσταση που θα απελευθέρωνε το πνεύμα, την οτροπία, τα μυαλά και τις αρχές εκείνες που όλους εμάς τους άνδρες και τις γυναίκες μας έβαλαν σε στεγανά, σε κλουβάκια, μας εγκλώβησαν σε κάποια στεγανά και έτσι μας απομόνωσαν όσον αφορά το μέλλον. Συμφωνίες λοιπόν που ε, είχαν ή δεν είχαν ε, υπογραφεί είναι μεν πολύ σημαντικές. Όμως πώς θα πρέπει να κινηθεί κανείς, πώς θα μπορεί η κοινωνία να κινηθεί προς ένα πιο ανοιχτό πλαίσιο προς ένα, μια πιο ανοιχτή προσέγγιση για τις γυναίκες, πιο δημοκρατική προσέγγιση και πώς θα μπορούσαμε να βρεθούμε ή σε ίση βάση και να αντιμετωπίσουμε τους Ισλαμιστές. Πώς να τους αντιμετωπίσουμε αυτούς και την συντηρητική κοινωνία που επί πολλά χρόνια δρούσαν. Πώς θα αντιμετωπίζαμε και θα μπορούσαμε να βρεθούμε απέναντι σε οποιαδήποτε εξουσία και στη στρατιωτική εξουσία που ήταν πολύ συντηρητική και είναι συντηρητική. Όλα αυτά είναι θέματα και ερωτήματα που μας απασχολούν. Να δούμε τι πρέπει να κάνουμε εμείς γυναίκες και άντρες. Γιατί δεν είμαστε μόνο οι γυναίκες που υποφέραμε υπό, αυτές, υπό αυτά τα δικτατορικά καθεστώτα επί δεκαετίες. Και οι άντρες και οι γυναίκες υπέφεραν πήραμε και παίρναμε τον πρωτοπόρο ρόλο προπομπή κατά τα τελευταία αυτά χρόνια διότι θεωρήσαμε ότι δεν θα μπορούσαμε αμέσως να καταλήξουμε σε φυλακές όπως οι άντρες που θα συλλαμβανόντουσαν. Είχαμε λοιπόν το προτέρημα αυτό του να είμαστε εντός εισαγωγικών δεύτερης κατηγορίας πολίτες, ακόμα και στην καταστολή, στην καταπίεση. Οι πρώτα καταπιεζόντουσαν και διοκόντουσαν οι άντρες και μετά εμείς. Αλλά μια και έγινε και ξέσπασε η Επανάσταση, από τότε που ξέσπασε οι γυναίκες ήταν η αιχμή του δόρατος. Η αιχμή του δόρατος της Επανάστασης. Η, εμ, εμπροστοφυλακή. Και τώρα έχουμε μια ολόκληρη ομάδα, ένα πυρήνα που συνεχίζει να δρά και συνεχίζει τη δράση, του ο πυρήνας αυτός με ιδιαίτερο σθένος ε, κατά της ε, στρατιωτικής εξουσίας. Αυτές, η, αυτή η ομάδα είναι όλες γυναίκες, νέες γυναίκες, σύγχρονες γυναίκες που βρίσκονται δίπλα σε άντρες, δίπλα στους άντρες ζητούν αμέσως να σταματήσουν οι στρατιωτικές δίκες στα στρατοδικεία και αυτή τη στιγμή τέσσερις ή πέντε γυναίκες έχουν συλληφθεί μέχρι σήμερα και έχουν προσαχθεί στα δικαστήρια για να δικαστούν και καταδικαστούν. Είναι ενδιαφέρον να δει και να γνωρίζει κανείς ότι η πορεία και η μετάβαση από τις πλατείες όπου διαδηλώσαμε, διαδηλώναμε και ζήσαμε, βιώσαμε αυτή την επανάσταση και το κοινοβούλιο και πώς μηχανή, οι πολιτικοί μηχανισμοί λειτουργούν. Είναι πολύ ενδιαφέρον να το δει κανείς. Για πρώτη φορά οι γυναίκες συμμετέχουν σε τέτοιο ευρύ πλαίσιο και βαθμό. Πολιτικά κόμματα που υιοθετούσαν τις ίδιες μεθόδους όπως το παλαιό καθεστώς βάζοντας τις γυναίκες στο περιθώριο, τώρα βλέπουμε ότι προσκαλούν τις γυναίκες να συμμετάσχουν και ενδιαφέρονται οι γυναίκες να διαδραματίσουν ένα σημαντικό, πολύ σημαντικό ρόλο. Θέλω να σας πω ότι τις επόμενες εβδομάδες θα δούμε και θα βρούμε τις γυναίκες και τους άντρες να εμένουν και να επιμένουν και να ασκούν πίεση. Πρώτα να υιοθετηθεί και να εγκριθεί το Σύνταγμα και αυτό να έχει πρωτεύοντα ρόλο έναντι των στρατιωτικών αρχών ή του στρατιωτικού συμβουλίου που είπαν πρώτα να γίνουν λέει εκλογές και μετά να υιοθετηθεί Σύνταγμα. Θέλω να σας πω στις επόμενες εκλογές που θα γίνουν το Σεπτέμβριο 2011 θα ασκήσουμε πίεση να αναβληθούν αυτές οι εκλογές, να έχουμε περισσότερο χρόνο να διοργανωθούμε, να να υιοθετήσουμε ένα σύνταγμα το οποίο θα είναι το καλύτερο δυνατόν για το μέλλον της χώρας μας, αυτής της χώρας μας. Και εν τέλει, τέλος, θέλω να σας πω ότι το κοινοβούλιο το οποίο θα συγκροτηθεί δεν θα έχει με ποσόστοση γυναίκες όπως είχε το τελευταίο μας κοινοβούλιο, διότι πιστεύουμε ότι από τότε που βρισκόμαστε εμείς επικεφαλής πλέον ως γυναίκες δεν χρειάζεται μία θετική ε, διακριτική μεταχείριση έναντι της αρνητικής διακριτικής μεταχείρισης που υφίστατο στο παρελθόν και έτσι βλέποντας ότι ε, έχει, το παλαιό καθεστώς είχε κάποιες νέες ε, βλέψεις και ότι υπήρχαν οποιοδήποτε παράδειγμα Ισλαμιστές ε, που αν θα τολμούσαν να μειώσουν σε οποιοδήποτε βαθμό την, το βαθμό της ελευθερίας των Αιγυπτίων θα έπρεπε να πληγούν άμεσα. Θα είμαστε εμείς που θα δώσουμε αυτόν τον αγώνα. Ευχαριστώ. σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας αυτή και για την παρουσίασή σας του ρόλου ρόλου των γυναικών και της κατάστασης των γυναικών στην Αίγυπτο. Τώρα θα ήθελα να δω, υπάρχουν κάποιες παρεμβάσεις για ερωτήσεις προς ε, τις ε, όσες εξεφώνησαν λόγους και παρενέβησαν. Εσείς παρακαλώ κυρία. Ευχαριστώ για την συνάντηση αυτή. Ευχαριστώ για τις εξαιρετικές παρεμβάσεις που μας ευνοούν όλους Μία ερώτηση για την κυρία Σμάιλ για την κατάσταση στην Αίγυπτο. Υπάρχει ένας μεγάλος συνασπισμός με φιλελεύθερα κόμματα, με σαλαφιστικά κόμματα και με, με την Ισλαμική αδελφότητα, με τους μουσουλμάνους αδελφούς μάλλον. Δεν το καταλαβαίνουμε αυτό. Τι σημαίνει αυτό ιδιαίτερα για το μέλλον των γυναικών. Πώς μπορεί κανείς να διασφαλίσει τα συμφέροντα των γυναικών μέσα από έναν τόσο ευρύτατο συνασπισμό που κάποιοι εταίροι ακολουθούν θρησκευτικές πεπιθήσεις περιοριστικές για το ρόλο της γυναίκας στην οργάνωση του κράτους και ε, ένα πιθανώς μη θρησκευτικό σύνταγμα. Θα μαζέψω αρκετές ε, πρώτα ερωτήσεις και μετά θα μπορέσετε να απαντήσετε. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που οργανώνει αυτήν την συνάντηση για να δώσει το λόγο στις γυναίκες. Η ερώτησή μου είναι προς την κυρία Ισμαέλ. Είπατε στην παρέμβασή σας ότι οι γυναίκες της Αιγύπτου δεν θα έχουν ανάγκη από ποσοστώσεις για να πετύχουν να κατακτήσουν τα δικαιώματα που τους αναλογούν και ότι θα ανταποκριθεί ο Αιγυπτιακός λαός. Στο Αιγυπτιακό σύστημα προβλέπονται ποσοστώσεις για τις επόμενες εκλογές. Ευχαριστώ. Μια ερώτηση για την κυρία Ελγκάλη. Μπορείτε να περιγράψετε τον ρόλο σας σε αυτό το νέο προσωρινό συμβούλιο. Ποια είναι η θέση σας, τι ακριβώς κάνετε. Και μια δεύτερη ερώτηση είναι ότι ακούμε πολλά για σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Θα θέλαμε να μας δώσετε περισσότερες εξηγήσεις Και μία ερώτηση για την κυρία Ζουίνη. Η νέα πολιτική γειτονία στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα βασίζεται στο υπόλογο και των δύο πλευρών και στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλο και περισσότερο. Τουλάχιστον αυτός είναι ο στόχος. Πιστεύετε ότι μπορούμε εμείς να ζητήσουμε η κατάσταση των γυναικών να είναι ένα από τα κριτήρια αξιολόγησης της κατάστασης και πιστεύετε ότι και για το δικό σας κίνημα ένα μια τέτοια κίνηση θα είναι κάτι το χρήσιμο. Καλώς. Λοιπόν, θα ήθελα να δώσω το λόγο στις τρεις ομιλήτριες για να περάσουμε στο δεύτερο πάνελ αμέσως μετά. Αρχίζουμε ανάποδα τώρα με τη σειρά ομιλίας η κυρία Ισμαήλ Σχετικά με το συνασπισμό των πολιτικών. Έχουμε τρεις μεγάλες πολιτικές συμμαχίες. Ε, μία από αυτές είναι μεγαλύτερη ομπρέλα θα έλεγα που περιλαμβάνει πάρα πολλές πολιτικές δυνάμεις. Η οργάνωση πολιτική στην Αίγυπτο άργησε αργά Άρχισε λοιπόν πολύ αργά, χρειάστηκαν τρεις μήνες μέχρι τις αρχές Μαΐου για να εκπροσωπηθούν όλοι, εκτός από τους Ισλαμιστές οι οποίοι δεν δέχτηκαν να συμμετέχουν. Βέβαια σε μια ιστερότερη φάση και οι Ισλαμιστές θα πάρουν μέρος. Έχουμε σαν στόχο δύο πράγματα. Πρώτον, να δημιουργήσουμε μια μεγάλη ομάδα υποψηφίων που θα κατέλθουν για να καταπολεμήσουν τις ιδέες και τις αντιλήψεις του παλαιού καθεστώσος, οι οποίες ιδέες θα είναι παρούσες εκεί και πολλοί θα κατέβουν στις εκλογές για την αποκατάσταση της παλιάς πολιτικής τάξης. Θέλουμε όλοι οι πολιτικοί να πάρουν μέρος στις διαδικασίες αυτές. Υπάρχουν επίσης δύο άλλες συμμαχίες ανάμεσα στα παλιά παραδοσιακά κόμματα και σε κάποιες κινήσεις της νεολαίας. Όλες αυτές οι συμμαχίες νομίζω ότι τελικά θα εξαρτηθούν από το αν θα υπάρξει μια συντριπτική θα έλεγα επικράτηση ε, μιας πολιτικής τάσης, είτε είναι οι Ισλαμιστές είτε όχι. Ακόμα και αν συμβεί κάτι τέτοιο δεν θα πρέπει να υπάρξει πανικός στον υπόλοιπο κόσμο, γιατί έχουμε φτάσει σε μια φάση πλέον όπου οι Αιγύπτιοι ε, θα αντισταθούν εναντίον Ιουδήποτε ο οποίος θέλει να τους επιστρέψει σε καθεστώς ανελευθερίας ακόμα και αν είναι θρησκευτικές δυνάμεις αυτές σχετικά με τις ποσοστώσεις. Δεν είναι τίποτα ξεκάθαρο ακόμα, αλλά από ό,τι γνωρίζουμε δεν θα υπάρξουν ποσοστώσεις για τις γυναίκες στο επόμενο κοινοβούλιο. Υπήρχαν ποσοστώσεις το 2010 στις κοινοβουλευτικές εκλογές και εγώ ήμουνα εκτός των ποσοστώσεων υποψήφια γιατί είχε σαν στόχο να δώσει στις γυναίκες περισσότερες έδρες. Λοιπόν, έδινα στις γυναίκες λουλούδια για να ψηφίσουν το κυβερνόν κόμμα τότε, αλλά τις γυναίκες του κυβερνόντος κόμματος. Σε βάση περιπτώσει δεν θα υπάρξουν μάλλον ποσοστώσεις για την επόμενη Βουλή. Ελπίζουμε όμως τελικά το Σύνταγμα να σέβεται τις προσωπικές ελευθερίες όσο περισσότερο γίνεται γιατί και πολλοί συνάδελφοι πολιτικοί στην Αίγυπτο θεωρούν ότι οι προσωπικές ελευθερίες και ο σεβασμός των προσωπικών ελευθεριών είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό για την ολοκλήρωση της Επανάστασης. Το θέμα δεν είναι να απομακρύνεις μία μορφή εξουσίας και να την αντικαταστήσεις με μία άλλη, αλλά να την αντικαταστήσεις με τον σεβασμό των δικαιωμάτων σου και των αξιών σου. Σας ευχαριστούμε. Αν κατανόησα σωστά, υπάρχει ένα συνασπισμός των παλαιών ε, κομμάτων, είπατε και ένας από αυτούς τους συνασπισμούς ε, έχει τους ε, μουσουλμάνους αδερφούς που δημιουργήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα και υποστηρίζεται από 12 παραδοσιακά κόμματα και τους μουσουλμάνους αδερφούς. Η άλλη αυτή η ένωση δεν έχει τους μουσουλμάνους αδελφούς αλλά νομίζω θα συμμετάσχει και οι εκλογές θέλουμε, παλεύουμε να αναβληθούν και άλλες συνασπισμοί που είναι μικρότεροι και έχουν και κάποια νέα κόμματα, αποκοινούμε κάποια παλαιά, ουσιαστικά όλοι προσπαθούν να δημιουργήσουν τα θεμέλια και τη βάση για μια κοινωνία των πολιτών που θα σέβεται τα, τα πολιτικά δικαιώματα. Σας ευχαριστούμε για αυτή την αποσαφήνιση, για αυτή τη διευκρίνηση. Και όπως είπατε, είσαστε πολύ αισιόδοξοι όπως αναφέρθηκε και ελπίζω μπορούμε να συμμετάσχουμε σε αυτή την αισιοδοξία για τον ρόλο των γυναικών που είχαν ενεργοποιηθεί ενεργά σε αυτή την ε, επανάσταση. Και Ελπίζουμε ότι ο αγώνας σας για τα δικαιώματα του ανθρώπου θα είναι και μια προσπάθεια για τα δικαιώματα των γυναικών και τα δημοκρατικά τους δικαιώματα. Οι επιφυλάξεις που έχουμε για την Συνταγματική Επιτροπή ουσιαστικά ξεπερνούν την εκπροσώπηση των γυναικών ως θέμα φίλου σε αυτή την Επιτροπή. Είχαμε επιφυλάξεις όσον αφορά τις πολιτικές τάσεις και τις θρησκευτικέ τάσεις κάποιων μελών. Είχαμε επιφυλάξεις κατά του γεγονότος ότι εκ των άνω ξεκινούσε και ήθελε να επιβληθεί. Εμείς θέλαμε να επιλέξουμε τα μέλη αυτής της Επιτροπής. Δεν έχουμε καμιά αντίρρηση να είναι όλοι άνδρες ή όλοι γυναίκες εφόσον θα εκπροσωπεί την πλειοψηφία των επαναστατών για το τι θεωρούν ότι ποια μορφή θα πρέπει να πάρει το Σύνταγμα. Ευχαριστώ. Και θα δώσω τώρα την Προεδρία στον λόγο με συγχωρείτε, εξ αριστερών δεν ξέρω ποια θα ήθελε να παρέμβει πρώτη. είναι, είπατε ποιος είναι ο ρόλος μας στο ε, Συμβούλιο Μετάβασης. Εκπροσωπώ τη Βεγγάζη. Είμαι επίσης πρόεδρος της Νομοθετικής Επιτροπής του Συμβουλίου. Όταν ανέλαβα αυτή την θέση της Προέδρου της Νομικής Επιτροπής δημιουργήσαμε υποεπιτροπές οι οποίες θα ασχοληθούν με τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν με την Επανάσταση. πιο σημαντική από αυτές τις υποεπιτροπές ασχολείται με τη συλλογή αποδείξεων για τα εγκλήματα του καθεστώτος και συνεργάζεται με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και παρέχει όλες τις απαραίτητες ενδείξεις και αποδείξεις για να αποκαλυφθούν τα εγκλήματα και να υποστηριχθεί προσφυγή στο Διεθνές Ποινικό σήμερα. Στόχος μας λοιπόν είναι η συλλογή αποδείξεων και για την ύπαρξη μισθοφόρων και φυλακισμένων τους οποίους χρησιμοποιεί ο Καντάφη για να κυνηγήσει και να καταπολεμήσει τον Λιβικό λαό. Συλλέγουμε πληροφορίες για τον αριθμό του, συντονίζουμε τις προσπάθειές μας με τις διεθνείς ΜΚΟ που έρχονται στην Λιβύη και εξετάζουν τους φιλοξενούμενους και τους μισθοφόρους. Το προσωρινό συμβούλιο επέτρεψε από την πρώτη στιγμή της ύπαρξής του στον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό, στο Human Rights Watch και στις διάφορες ΜΚΟ να κάνουν έρευνες ε, με, για τους ε, φυλακισμένους, ε, τους εχμαλώτους κτλ. Και δεν εμποδίσαμε κανένα να έλθει στη χώρα. Η Τρίτη Επιτροπή ασχολείται με την προετοιμασία των σχεδίων νόμου που απαιτούνται ε, να είναι σε θέση λειτουργίας πλέον στην επόμενη φάση. Είπαμε ότι η Λιβύη δεν είχε σύνταγμα για 42 χρόνια. Σήμερα έχουμε την ανάγκη να έχουμε νέους νόμους που να ρυθμίζουν και να οργανώνουν την μεταβατική περίοδο μετά την πτώση του Γκαντάφη. Δεν έχουμε εκλογικό νόμο, δεν έχουμε νόμο ε, για δημοψήφισμα Προσπαθούμε λοιπόν να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να οργανώσουμε τις εκλογές. Η εργασία, Η εργασία της Επιτροπής οδήγησε στην ε, κατάρτιση ενός ε, καταστατικού ε, χάρτη για να δούμε ποια είναι τα συγκεκριμένα βήματα που θα ζήσει η Λιβύη μετά την πτώση του δικτάτορα. Πρώτο θέμα. Δεύτερο το θέμα του βιασμού και της σεξουαλικής βίας. Από τους ε, μπάτσους ε, του Καντάφη. Δυστυχώς ακόμα δεν έχουμε συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία και στατιστικές στον τομέα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να γνωρίζει κανένα την αλήθεια σε μια ανατολίτικη κοινωνία με τις ιδιαιτερότητες του πολιτισμού μου. Δεν μπορούμε να έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία. Υιοθετήσαμε λοιπόν τη μέθοδο των ερωτηματολογίων. Προσπαθούμε να συλλέξουμε κατά τι περισσότερες ε, πληροφορίες. Αλλά οι γυναίκες δεν θέλουν να απαντήσουν γιατί φοβούνται την αντίδραση τη κοινωνίας όταν γίνει γνωστή η κατάστασή του το πάθος του δηλαδή. Δεν έχουμε λοιπόν συγκεκριμένε στατιστικέ. Ξέρουμε ότι είναι πολύ διευρυμένο αυτό το έγκλημα, αλλά είναι πολύ δύσκολο να το αντιμετωπίσουμε λόγω του πολύ λεπτού χαρακτήρα του μέσα στην κοινωνία μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για τις ευκρινήσεις. Εγώ έχω μία ερώτηση. Σας γρήγορα όταν είπατε για την σύνταξη του συνταγματικού κειμένου. Κατά πόσο θα συμπεριλάβετε εκεί τα δικαιώματα των γυναικών. Είναι ένα βασικό θέμα. Μπορείτε να μας περιγράψετε κάτι σχετικά. Ε, δεν είναι σύνταγμα δεν είναι σύνταγμα αυτό μπορούμε να το ονομάσουμε ίσως μεταβατικό σύνταγμα για να οργανωθεί η ενδιάμεση περίοδος περιμένοντας ε, την διατύπωση ενός πραγματικού συντάγματος. Δεν θα είναι αυτό το σύνταγμα της χώρας. Σχετικά με αυτή τη χάρτα λοιπόν, την οποία επεξεργαζόμαστε, πράγματι περιλαμβάνει ε, κάποια στοιχεία για τα δικαιώματα των γυναικών και των ανδρών φυσικά, και νομίζω ότι δεν θα είναι όμως το τελικό σύνταγμα της χώρας. Το μελλοντικό σύνταγμα προφανώς και θα υπάρχουν ρυθμίσεις οι οποίες θα καθιερώνουν τα δικαιώματα των παιδιών και των γυναικών. Ευχαριστώ πολύ για τις διαφημίσεις σας. Νομίζω ότι η επαναστατική διαδικασία αυτός είναι ο σωστός όρος. Δεν έχει πετύχει ακόμα τους στόχους της. Βρισκόμαστε σε μια επαναστατική διαδικασία η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και κάποια χρόνια, η οποία όμως τώρα εξελίσσεται λόγω ακριβώς ε, του επίπεδου ε, της συνειδητοποίησης των πολιτών στην Τινησία. Πρέπει να κατανοήσουμε αυτή την επαναστατική διαδικασία. Αυτή η διαδικασία, αυτή η αλλαγή στην Τινησία δεν είναι μήνυμα μόνο για όλη την περιοχή, αλλά θα πρέπει το μήνυμα αυτό να φτάσει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί τον τελευταίο καιρό η Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι την τελευταία στιγμή έδινε ε, προτιμησιακές συμπεριφορές στον ε, δικτάτορα Μπεν Αλή, υποστηριζόταν πλήρως από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να σας πω την αλήθεια, ακόμα και αν είναι δυσάρεστη, θα έπρεπε το Κοινοβούλιο και τα ευρωπαϊκά όργανα να δουν πράγματι ποια είναι τα κριτήρια με τα οποία υποστηρίζονται διάφορα καθεστώτα και όχι μόνο τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είπατε ότι το άρθρο 2 της Συμφωνίας της Βαρκελόνης, της Σύμβασης της Βαρκελόνης, ποτέ δεν, δεν έγινε αντικείμενο σεβασμού από τον Πεναλή και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε πάντα τα στραβά μάτια και τα ανθρώπινα δικαιώματα ποτέ δεν έγιναν πλήρως σεβαστά από τις χώρες που υπέγραψαν αυτές τις συμφωνίες, ποτέ δεν πιέστηκαν τα καθεστώτα Ίσως αυτές οι νέες δημοκρατικές χώρες, αυτές οι αναδυόμενες δημοκρατίες να δώσουν την απάντηση και τα νέα κριτήρια που θα πρέπει να υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ίσως θα πρέπει να δείξουμε και μια κάποια ταπεινοφροσύνη απέναντι σε αυτούς τους λαούς που πολλά είναι ικανοί να κάμνουν. Φυσικά πολλά θα εξαρτηθούν από το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά εμείς οι γυναίκες σαν φεμινίστριες στην Ισία είμαστε υπόλογες και για την εικόνα της γυναίκας στη δημόσια σκηνή, αλλά και για την υιοθέτηση κανόνων και νόμων για τις γυναίκες που να είναι εναρμονισμένοι με τις διεθνείς συμβάσεις ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το λέω αυτό γιατί όλα τα πολιτικά κόμματα τώρα είναι υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών και θεωρούν τα κεκτημένα των γυναικών δεδομένα. Ξέρετε ότι έχουμε ένα προσωπικό κώδικα πολύ προχωρημένο. Αυτό σημαίνει ότι η ισιακή κοινωνία έχει ήδη ενσεματώσει το ότι τα κεκτημένα αυτά είναι τμήμα της πολιτιστικής ε, προέλευσης των Τινησίων. Ακόμα και τα Ισλαμικά κόμματα αναγνωρίζουν την κατάσταση αυτή Παρ' όλα αυτά είμαστε πολύ επιφυλακτικές. Ξέρουμε ότι μιλάμε για προεκλογικές εκστρατείες. Είμαστε πάρα πολύ προσεκτικές. Βλέπουμε όμως ότι σήμερα, εν πάση περιπτώσει, τα δικαιώματα των γυναικών είναι τμήμα των προγραμμάτων των πολιτικών των πολιτικών κομμάτων και όλα λένε ότι θέλουν να σεβαστούν τον κώδικα αυτά και κανένας πολιτικό σχηματισμός δεν αμφισβητεί τα δεδομένα και τα κεκτημένα των ε, ισίων γυναικών. Εμείς δεν θέλουμε να μείνουμε στα κεκτημένα, θέλουμε να περάσουμε προς την ουσιαστική ισότητα και θέλουμε ουσιαστική αυτή η ισότητα να αναφέρεται στο Σύνταγμα, όχι μόνο σε επίπεδο αρχής, αλλά και στα πλαίσια και της διαδικασίας για την καταπολέμηση των διακρίσεων και του δικαιώματος της αξιοπρέπειας. Πώς να επιβάλλουμε λοιπόν στο νέο σύνταγμα έτσι να λαμβάνει υπόψη ε, και τις γυναίκες και τους άνδρες ε, να μπει και η αναφορά στις γυναίκες ξεκάθαρα στο Σύνταγμα να αναφέρεται στους πολίτες άνδρες και γυναίκες και την καταπολέμηση των διακρίσεων για λόγους φιλετικούς, για λόγους θρησκευτικού κτλ. κτλ. Πιστεύουμε ότι η αρχή της μη διάκρισης είναι μια διαδικασία πολύτιμη που λαμβάνει υπόψη όχι μόνο σε επίπεδο αρχής την ισότητα γιατί μπορεί να λέμε ναι στην ισότητα αλλά όταν μιλάμε για την καταπολέμηση των διακρίσεων τότε είναι πιο αποτελεσματική η παρέμβασή μας. Ε, Θαυμάσια. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Μία ερώτηση ακόμα. Και μετά πρέπει να ολοκληρώσουμε εδώ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Έχω μια ερώτηση όπου δεν γνωρίζω αν είναι σε θέση να απαντηθεί από τις συμμετέχουσες, αλλά με απασχολεί αυτό το ερώτημα. Εμείς στο τέλος ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να εγκρίνουμε ή να μην εγκρίνουμε τη διμερή συμφωνία εμπορίου με το Μαρόκο. Και όταν έχουμε το θέμα των δικαιωμάτων των γυναικών και τα συζητούμε αυτά, φυσικά είναι σημαντικά σημεία αυτά, αλλά στο τέλος πρέπει να είναι δυνατόν οι γυναίκες να συμμετάσχουν στην οικονομική ζωή με τον ίδιο τρόπο και στον ίδιο βαθμό όπως και οι άντρες και, αν, και όταν έρχεται η ώρα και έρθει η ώρα να συζητήσουμε για αυτή την εμπορική συμφωνία με το Μαρόκο, είναι ένα θέμα αυτό για μένα. Εποφελείται ο πληθυσμός της χώρας αυτής. Εποφελούνται οι πολίτες, οι εργαζόμενοι, η παραγωγή για παράδειγμα των γεωργικών προϊόντων. Σε αυτή τη χώρα εποφελούνται από αυτή τη συμφωνία ή συνάπτουμε εμείς μια συμφωνία που εξυπηρετεί μεγάλες επιχειρήσεις μόνο και τα συμφέροντά τους. Δεν ξέρω αν είσαστε σε θέση να απαντήσετε αυτή την ερώτηση. Θα με ενδιαφέρε πάρα πολύ να απαντηθεί όμως. Ευχαριστώ. Ίσως η κυρία Μπατρούι να μπορέσει να απαντήσει. Ε, Δεν ξέρω αν η κυρία Βουλευτή γνωρίζει το σχέδιο ενός νέου συντάγματος στο Μαρόκο που ε, παρουσίασε η, αυτή τη ε, στις 17 Ιουνίου προχτές κατά διάρκεια ακριβώς ε, όπως ανέφερε η κυρία Βουλευτής ε, τα δικαιώματα γυναικών ε, αυτό το σχέδιο συντάγματος αναφέρεται στην ισότητα ανδρών και γυναικών σε όλους τους τομείς οικονομικούς, κοινωνικούς, περιβαλλοντολογικούς, οικονομικούς και ούτω καθεξής. Εκτός αυτού προστίθεται στο κείμενο Να το βρω στο έγγραφό μου εδώ. Η ισότητα, όπως σας είπα, ναι. Όπως είναι το κείμενο της Ευρωπαϊκής που υπευλήθη για το σχέδιο του συντάγματος, επί βάσης ισότητας ανδρών γυναικών τα πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά, πολιτιστικά κοινότητα, επίσης η δημιουργία ενός μηχανισμού ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Αυτό είναι το σχέδιο συντάγματος, για το οποίο θα πρέπει να ψηφίσουν την 1η Ιουλίου οι Μαροκινοί και που θα αλλάξει φαντάζομαι πολλά στην κοινωνία μας. Όσον αφορά το δεύτερο ερώτηση, κατά πόσον οι εργαζόμενοι σε όλες τις ε, περιοχές του Βασιλείου μπορούν να αφοληθούν από τις ε, εμπορικές συμφωνίες. Δεν μπορώ πραγματικά να, αποφάσω, να απαντήσω άμεσα. Αλλά εάν οι ομάδες που εκπροσωπούν την μαροκινή οικονομία ωφεληθούν, αυτές οι μεγάλες ε, ομάδες, οι επιχειρήσεις ε, θα μπορέσουν να βοηθήσουν όλους τους Μαροκινούς, κατά την γνώμη μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα έχετε ίσως περισσότερες να συζητήσετε στο επόμενο πάνελ το θέμα αυτό. Εκτός αν κάποιος άλλος θέλει να απαντήσει. Πολύ σύντομα, όχι, ωραία, εντάξει. Είναι πολύ δύσκολη η ερώτησή σα Το επόμενο πάνε, ίσω θα σα δώσω περισσότερε απαντήσει. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους που συμμετείχαν εδώ. Παρακαλώ να παραμένετε μαζί σας. Θα αλλάξουμε εδώ το πάνελ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους ομιλητές που πήραν το λόγο και να σας ευχαριστήσω κάθε επιτυχία στις μάχες που έχετε ακόμα να δώσετε. Αν υπάρχει κάτι που πιστεύετε θα πρέπει να γνωρίσει το Κοινοβούλιο, παρακαλώ ενημερώστε μας. Και κρατήστε την, το κουράγιο σας, την δύναμή σας. Πολλά κάνετε για μας γυναίκες. Ευχαριστώ. Παρακαλώ να ξεκινήσουμε με τον επόμενο γύρο. Εκείνοι που επιθυμούν να παραμείνουν στην αίθουσα μπορούν να παραμείνουν. Εκείνοι που θέλουν να συζητήσουν παρακαλώ να αποχωρήσουν. Αυτό θα ήταν πολύ χρήσιμο αν γινόταν. Παρακαλώ λοιπόν. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, My name is Michael είναι το όνομά Θα, προεδρεύω στο τελευταίο τμήμα αυτή τη συνεδρίαση. Είμαι της Επιτροπής Ανάπτυξης, Ήμουν Ευρωβουλευτής για περίπου 12 χρόνια. Είμαι Ευρωβουλευτή και είμαι επίση ε, και στην Επιτροπή ε, για θέματα δικαιοσύνης εσωτερικών και σε σχέση με την διακομματική ομάδα για τους ομοφιλόφιλους και τους ε, transsexuals. Είναι σημαντικό οι γυναίκες ε, να είναι πλειοψηφία που είναι πλειοψηφία. Κάνουμε λόγο για μειονότητες ε, στην Ευρωβουλή και χαίρομαι στο να πω ότι ανήκω εγώ σε μία από αυτές τις μειονότητες. Είμαι ομοφιλόφιλος, ανοιχτά ομοφιλόφιλος και γι' αυτό λοιπόν γνωρίζω και έχω συνειδητοποιήσει πάρα πολύ καλά την αρνητική διακριτική μεταχείριση που βιώνουν καθημερινά όσοι είναι, ανήκουν σε αυτή τη μειονότητα καθημερινά στη ζωή τους. Διερωτώνται κάποιοι και λένε τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για τις χώρες της Βόρειας Αφρικής, της Μέσης Ανατολής και πέρα από αυτές. Ε, τι μπορούμε να κάνουμε. Είναι ενδιαφέρον ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορούν να κάνουν πάρα πολλά πράγματα, μπορούν να πράξουν. Πολλά έγινε έγιναν πρόσφατα. Αλλά πολλά περισσότερα ακόμα απομένουν και πρέπει να γίνουν. Έχουμε τα μέσα, τα εργαλεία να προασπιστούμε, να υπερασπιστούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των γυναικών και τα δικαιώματα των ομοφιλοφίλων και των transsexual, τα δικαιώματα όσον αφορά τα συνειδησιακά δικαιώματα και την ελευθερία συνείδησης. Όλα αυτά είναι δικαιώματα που ε, κατοχυρώνονται στις αρχές και τις αξίες της συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ιδρυτική συνθήκη της Ρώμης και και οι επακόλουθες συνθήκες σε αυτά βασίζονται και η συνθήκη του Αμστερντάμ και πρόσφατα η συνθήκη της Λισαβόνας. Έχουμε συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου με πάρα πολλές χώρες και το άρθρο 2 αυτών των, ελευθέρων, των ε, συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου είναι η προαγωγή και η υπεράσπιση, η προάσπιση των ε, δικαιωμάτων του ανθρώπου, των δικαιωμάτων ε, της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Όμως υπάρχουν διαρκώς παραβιάσεις αυτών των δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των γυναικών και έχουμε αποτύχει στο να δρομολογήσουμε δράση υπό το άρθρο 2. Μόνο μία φορά υπεψήφισε το πάγωμα το Ευρωκοινοβούλιο μιας Ευρωπαϊκής Συμφωνίας Εμπορίου. Ήταν η Συμφωνία Εμπορίου με το Ισραήλ και το Συμβούλιο και τα κράτη-μέλη δεν δραστηριοποιήθηκαν σε σχέση με αυτή τη σύσταση του Ευρωκοινοβουλίου. Έχουμε και τη Συμφωνία Κοτονού και έχουμε συμφωνίες ε, με όλες τις χώρες ΑΚΕ της, ε, ε, του Ειρηνικού, της Καραϊβικής, της Αφρικής και όλα αυτά υπογραμμίζουν τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πάλι στην διαπραγμάτευση μια τέτοια ε, συμφωνία ε, εδώ και ε, λίγου μήνε πριν η αντίσταση των χωρών και της Αφρική Καραϊβική και του Ειρηνικού όπου και όταν υπάρχουν θέματα παραβιάσεων και αγνόησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπήρχε αντίσταση, υπήρχε, υπήρχαν τριβέ και δεν κατέληξαν στο να συμφωνήσουν, στο να επιβληθεί αυτό ακριβώ το άρθρο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τι πολιτικέ ελευθερίε. Υπάρχει λοιπόν υπάρχουν αντιστάσεις όπως πολύ συχνά συμβαίνει. Η μία μειονότητα αποτελεί πιόνι στο παιχνίδι ε, εναντίον μιας άλλης μειονότητας. Σε αυτή τη συνάντηση, αυτή η συνεδρίαση αφορά τον ρόλο των γυναικών και οι γυναίκες πάντα ήταν προπομπή, πρωτοπόροι στον αγώνα και στις μάχες για τη δημοκρατία, κάνοντας δουλειά στα παρασκήνια πολλές φορές, χρησιμοποιώντας ε, και δίκτυα. Και αν δούμε τη δουλειά που έγινε στην Τινησία, στην Αίγυπτο, στο Μπαχρέιν, τη Σαουδική Αραβία όπου πρόσφατα 29 γυναίκες είχαν το θάρρος να προκαλέσουν την, σε σχέση με αυτή τη γελία απαγόρευση, αυτή την απαράδεκτη απαγόρευση να μην μπορούν να οδηγούν αυτοκίνητα οι γυναίκες αν έχουν κιόλας δίπλωμα οδήγησης. Είναι άτομα σαν αυτές τις γυναίκες που αλλάζουν τον κόσμο στον οποίο ζούμε και για να υπάρξουν αυτέ οι αλλαγέ πρέπει να βεβαιώσουμε ότι αυτέ οι αλλαγέ θα κατοχυρωθούν και θα ενταχθούν στο νόμο και με νόμιμε και νομικέ διαδικασίε και νομοθετήματα και γι' αυτό είμαστε υπερήφανοι για το ότι έχουμε ω Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα νομικά και ε, οικονομικά και μέσω των συμφωνιών μα για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα ώστε να είμαστε αποτελεσματικοί στου στόχου μα. και σε σχέση με αυτά τα οποία ο πρόεδρος Μπαρόζος στις 2 Μαρτίου σε σχέση με την, ε, ε, τα κονδύλια για την, ε, που εγκρίνονται όσον αφορά την εξωτερική δράση και τη βαρώνει άστον και τόσες πολλές δράσεις που αναλαμβάνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα ήρθε η χρονική στιγμή να δούμε το θέμα του καθεστώτος των γυναικών ως θέμα με σημασία, ιδιαίτερη σημασία, σημασία κλειδιού για τις χώρες αυτές. Και επιτρέψτε μου να αναφέρω παράθεμα από την ιστοσελίδα οι ανισότητες όσον αφορά το φύλλο είναι ένα από τα πιο σοβαρά προσκόμματα όσον αφορά την ανάπτυξη των ανθρώπων, του ανθρώπινου δυναμικού στις αραβικές χώρες. Μου λένε ότι το μικρόφωνο δεν λειτουργούσε. Λοιπόν, θα σας, υπο... σας υπόσχομαι ότι θα ξαναρχίσω από την αρχή. Η ισότητα των φύλων είναι ένα από τα πιο σημαντικά προσκόμματα και εμπόδια όσον αφορά τις αραβικές χώρες και βλέπουμε ότι και πέρα από τις αραβικές χώρες είναι ένα σημαντικότατο πρόσκομα παρόλες τις νομικές εγγυήσεις για τα δικαιώματα των γυναικών και τη συμμετοχή τους νομικά στην δημοκρατία υπάρχουν βαθιά ριζωμένοι ρόλοι ανδρών και γυναικών που είναι εμπόδιο στην πρόοδο αυτή και που υπάρχουν αυτά τα εμπόδια σε πολλές χώρες ε, του κόσμου. Έχουμε ε, προσκεκλημένους με τρεις ομιλητές. Η πρώτη είναι η Σοράια Μπαντάουι, που είναι η πρόεδρος ε, της Μαροκινής, του Μαροκινού Συλλόγου Επιχειρηματιών Γυναικών. Θα μας κάνει λόγο για τα βιώματά της και την πείρα της ως επιχειρηματία και κυρίως για το επιχειρήν και το πνεύμα το επιχειρηματικό στο Μαρόκο από τις γυναίκες σήμερα στο Μαρόκο. Έχει τον λόγο Σοράγια. Je Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Ένωση που δίνει τη δυνατότητα στις γυναίκες να ε, εκφραστούν σήμερα σε αυτήν την συνάντηση. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την πρόσκλησή σας. Χαίρομαι που είμαι εδώ στις Βρυξέλλες, πόλη όπου πέρασα ένα μεγάλο κομμάτι της νιώτης μου. Έχω ζήσει 16 χρόνια ε, ήμουν φοιτήτρια στις Βρυξέλλες και βρίσκομαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να μιλήσω για το ρόλο της γυναίκας και τη συνεισφορά της στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του Μαρόκου, της χώρας προέλευσής μου. Η ικανοποίησή μου είναι μεγάλη γιατί την πρώτη μου εμπειρία σαν γυναίκα υπεύθυνη επιχείρησης, επιχειρηματία, γεννήθηκε εδώ στις Βρυξέλλες. Ιστορία μιας επιτυχίας θα πούνε κάποιοι φίλοι, όπου ο άντρας μου και εγώ ξεκινήσαμε μια λυσίδα αρωματοπολίων στις Βρυξέλλες που κάποιοι από εσά σίγουρα έχουν επισκεφθεί. Το 1994 και ο άντρα μου και εγώ αποφασίσαμε να επιστρέψουμε στο Μαρόκο, δημιουργήσαμε μια νέα επιχείρηση, την Top Class Expresso που, μοιράζει, που διανέμει συγγνώμη, τους καφέδες Λαβάτσα και που είναι η επιχείρηση πιο σημαντική στον τομέα του καφέ στο Μαρόκο. Θα σας μιλήσω λοιπόν για τις επιχειρήσεις των γυναικών στο Μαρόκο, τον ρόλο της γυναίκας στην οικονομική ανάπτυξη και τον ρόλο της γυναίκας σε επίπεδο λήψεως αποφάσεων. Για να μπορέσει η γυναίκα να φτάσει σε αυτό το επίπεδο είμαι πεπισμένη ότι η εκπαίδευση είναι το βασικό στοιχείο, το βασικό χαρακτηριστικό που θα επιτρέψει στη γυναίκα να αποκτήσει τις απαραίτητες ικανότητες για να εξελιχθεί και να δημιουργήσει επιχειρήσεις σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας. Η Ένωση των Γυναικών Ηγετών Επιχειρήσεων στο Μαρόκο, της οποίας προεδρεύω, δημιουργήθηκε το Σεπτέμβριο του 2000 με τη βούληση μιας, ενός μικρού αριθμού γυναικών επιχειρηματιών που ήθελαν οι, φωνές τους, οι φωνές τους να ακουστούν. Παράλληλα με την προσπάθεια περιφερικοποίησης του Μαρόκου η παρουσία μας είναι δεδομένη σε, με 7 ε, τοπικές οργανώσεις και εκπροσωπούμε πάνω από 40.000 θέσεις απασχόλησης. Για να προωθηθεί η επιχειρηματικότητα των γυναικών, η ΑΦΕΜ, η, η οργάνωσή μας, συνεχίζει να προωθεί την εικόνα της γυναίκας επιχειρηματία που μπορεί να χρησιμεύσει σαν πρότυπο στις ε, υπόλοιπες γυναίκες και στις επερχόμενες γενιές. Στόχος μας είναι η προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας θέτοντας στη διάθεση των γυναικών τα απαιτούμενα μέσα για την ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους. Κατάρτιση, εκπαίδευση, δικτύωση Θέλουμε επίσης να ευαισθητοποιήσουμε τις γυναίκες σε διάφορους καινοτόμους τομείς. Κυρίες και κύριοι, όπως είπατε ήδη, οι στατιστικές δείχνουν ότι το ποσοστό των επιχειρήσεων στην περιοχή ΜΕΝΑ είναι από τους χαμηλότερους στον κόσμο, 16%. Συνειδητοποιώντας την κατάσταση αυτή και προσπαθώντας να τονώσουμε τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, Προσπαθούμε να προωθήσουμε κάποια προγράμματα που βελτιώνουν τη θέση της γυναίκας στο οικονομικό τομέα. Στόχος μας είναι να ξεπεράσει η γυναίκα τις δυσκολίες. Η γυναική επιχειρηματικότητα αντιμετωπίζει προβλήματα κοινωνικά, συνδυασμού ιδιωτικής και επαγγελματικής ζωής, δυσκολίας προσφυγής στη χρηματοδότηση, στα δίκτυα, στις αγορές, και να σας πω εδώ κάποια στατιστικά. Σύμφωνα με το Υπουργείο Προϋπολογισμού, η επιχειρηματικότητα των γυναικών το 2000 δεν ξεπερνούσε το 6,6% αλλά το 2004 φτάσαμε στο 10%. Υπήρξε λοιπόν μία πρόοδος τα τελευταία 10 χρόνια και σήμερα η επιχειρηματικότητα αντιπροσωπεύει το 12% των επιχειρήσεων. Παρ' όλα αυτά το αποτέλεσμα αυτό είναι πολύ πιο κάτω από τις προσδοκίες μας γιατί η γυναίκα αντιπροσωπεύει πάνω του 50% του πληθυσμού. Μια μεγαλύτερη εμπλοκή της γυναίκας στον τομέα τον επαγγελματικό θα επηρεάσει θετικά τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Η γυναίκα επιχειρηματία συνεχίζει να επενδύει στον τριτογενή τομέα και στον τομέα υψηλής τεχνολογίας. 60% των γυναικών είναι πτυχιούχοι πανεπιστημίου 70% είναι παντρεμένες και 77% περιορίζονται στις υπηρεσίες και στο εμπόριο στις μεγάλες πόλεις, 50% στον άξονα Καζαμπλάνκα Ραμπάτ. 57% είναι ανώνυμες εταιρείε και 22% προσωπικές. Αυτές οι τελευταίες είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις. 50% από αυτές έχουν κύκλο εργασιών κάτω των 5 εκατομμυρίων dirhams και πάνω του 65% έχουν προσωπικό χαμηλότερο από 19 πρόσωπα. Το ποσοστό θνησιμότητας είναι ιδιαίτερα ψηλό κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων χρόνων δημιουργίας των επιχειρήσεων. Η κατάσταση αυτή μας ανησύχησε. Προσπαθήσαμε εμείς να βελτιώσουμε τη δημιουργικότητα των γυναικών και το 2007 αναπτύξαμε ένα πρόγραμμα, το πρόγραμμα το εκολαπτήριο επιχειρηματιών, προσπαθώντας ε, να βοηθήσουμε τις γυναίκες να αντιμετωπίσουν επιμελητιακά τις ανάγκες τους. Προτείνουμε επίσης και διαφορετικά στάδια κατάρτισης, απόκτησης ικανοτήτων διαχειριστικών, σε συνεργασία με τα μέλη μας, έτσι ώστε να ενισχύσουμε τις επιχειρήσεις των γυναικών στη δύσκολη φάση της εκκίνησης. Βοηθήσαμε λοιπόν στην δημιουργία πάνω από 50 επιχειρήσεων σε διάφορους τομείς και 20 από αυτές έφυγαν από το λεγόμενο εκολαπτήριό μας και πετούν με τα δικά τους φτερά. Εμείς επαναλαμβάνουμε την εμπειρία αυτή και σε άλλες περιοχές του Μαρόκου. Ξεκινήσαμε με κολαπτήρια στο Ραμπάτ, στο Φες, στο Μαρακές, στην Ταγκέρι και γενιάσαμε μάλιστα το Φες την προηγούμενη εβδομάδα. Η επιτυχία των εκολαπτωμένων μας είναι η εγγύηση της αποτελεσματικότητάς μας. Οι στατιστικές του Υπουργείου Προϋπολογισμών δείχνουν ότι μειώθηκε ο αριθμός των εργαζομένων γυναικών τα δύο τελευταία χρόνια από 29% το 2005 σε 26% το 2010. Σύμφωνα με τις ίδιες στατιστικές το ποσοστό των νέων ανέργων είναι πολύ ψηλό, 25% στις γυναίκες, 17% στους άνδρες. Για να βοηθήσουμε λοιπόν την γυναίκα και την άνεργη γυναίκα ξεκινήσαμε το 2006 ένα άλλο πρόγραμμα το οποίο ονομάζουμε πρόγραμμα Reprofilage. Μια πρωτοβουλία για όλους τους πολίτες γιατί από τη μία βοηθούμε τις γυναίκες που έχουν δίπλωμα αλλά δεν έχουν θέση εργασίας με διάφορα στάζ, με διάφορες καταρτήσεις σε συνεργασία με τις ε, επιχειρήσεις που είναι μέλη της Ένωσής μας ε, βοηθάμε επίσης με προσωπικές οδηγίες τις ε, ε, γυναίκες αυτές για να παρουσιάζουν με σωστό τρόπο τις ικανότητές τους, την επαγγελματική τους επάρκεια και να τους διασφαλίσουμε την καλύτερη ένταξή τους στον χώρο των επιχειρήσεων. Μέσω αυτού του προγράμματος απαντάμε και στις προσδοκίες των μελών μας σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού. Μπορέσαμε μέσα από αυτή την εμπειρία να καταρτήσουμε άνω από 120 γυναίκες και 100 σχεδόν από αυτές έχουν ενταχθεί σε επιχειρήσεις. Για να ανακαλύψει κανείς λεπτομερώς το σύνολο των δράσεών μας που ελπίζουμε ε, ότι θα μπορέσουν να αναπτυχθούν και με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σας παραπέμπω στην ιστοσελίδα μας. αλφα. Από το 2011 οι αραβικές χώρες ε, της ε, Νότιας Μεσογείου βιώνουν λαϊκές εξεγεύσεις και έχουν αιτήματα για βαθιές μεταρρυθμίσεις. Και στο Μαρόκο ξεκινήσαμε σημαντικές μεταρρυθμίσεις από την αναρρίχηση στο θρόνο της μεγαλειότητάς του του Μωάμεφ του Έκτου. Θα αναφερθώ μόνο σε αυτές ε, στα πλαίσια του Μουνταουάνα, του κώδικα του αστικού του Μαρόκου που από το 2005 επιτρέπει στην ε, γυναίκα του Μαρόκου να είναι απόλυτα ισότιμη με τον άνδρα και ε, καθήρεσε ε, την έννοια του άνδρα κηδεμόνα. Είναι πρωτοποριακή η νομοθεσία αυτή στον αραβομουσουλμανικό κόσμο γιατί επιτρέπει στη γυναίκα να κατακτήσει τη θέση που της ανήκει στην κοινωνία. Πρόκειται για μια πραγματική επανάσταση του αστικού κώδικα που επιτρέπει στην γυναίκα να έχει λογαριασμό τραπεζικό, να δημιουργεί επιχειρήσεις, να ταξιδέψει εκτός του εδάφους του βασιλείου χωρίς γραπτή αδειοδότηση του άνδρα. Ο υπόλοιπος αραβομουσουλμανικός κόσμος δεν έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο ανεξαρτησίας. Ανάμεσα σε άλλα θετικά βήματα υπάρχει ο κώδικας εργασίας του 2004 σχετικά με τη συμμετοχή των γυναικών ε, στην εργασία και επίσης και η άδεια μητρότητας ε, που από 12 πήγε 14 εβδομάδες. και επίσης ίσχυσαν και αλλαγές σε σχέση με τη μετάδοση της υπηκότητας από τη μητέρα και όχι μόνο από τον πατέρα στα παιδιά. Στην ομιλία του στις 9 Μαρτίου η αυτού μεγαλειώτης προσκάλεσε όλες τις δόσες δυνάμεις της χώρας να συνεισφέρουν. Η Ένωσή μας όπως και άλλες προτάσεις καταθέσαμε τις προτάσεις μας για τη μεταρρύθμιση του συντάγματος διεκδικώντας την ισότητα ανδρών γυναικών στην ομιλία στις 17 Ιουνίου ή αυτού Μεγαλειώτης ανακοίνωσε το σχέδιο του νέου συντάγματος που λαμβάνει υπόψη και την φιλετική διάσταση ανακοινώνοντας την ισότητα του άνδρα και της γυναίκας για το αστικό δίκαιο σεβόμενη το σύνταγμα αλλά και τους νόμους που εμπνέονται από τη μουσουλμανική θρησκεία. Ταυτόχρονα αναγνωρίζονται ισότιμοι άνδρες και οι γυναίκες σε όλα τα πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά, πολιτιστικά και περιβαλλοντικά δικαιώματα και δημιουργείται μηχανισμός προώθησης της ισότητας ανάμεσα στον άνδρα και τη γυναίκα. Όλα αυτά τα είπε ο Βασιλιάς στις 17 Ιουνίου όταν εγκριθούν τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος την 1η Ιουλίου, τότε εμείς οι γυναίκες που παλεύουμε για την προώθηση του ρόλου της γυναίκας να κάνουμε κάθε προσπάθεια έτσι ώστε να επιτρέψουμε στις γυναίκες να προκόψουν στη χώρα μας συμμεριζόμενες στις καθολικές αξίες και στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πέρα από τις αλλαγές που έχουν ήδη γίνει, Υπάρχει μεγάλη προσπάθεια να περιμένουμε να υπάρξει μεγάλη προσπάθεια για να κερδίσει η γυναίκα τον χώρο που της αξίζει. Δεν ξέρω που είναι να σου πω την αλήθεια. Σας, παρακαλώ μπορείτε να τελειώνετε ε, γιατί δεν έχουμε τόσο χρόνο. Ναι η παρουσίαση μου είναι είναι μακρά, αλλά θα φτάσω στα συμπεράσματα ίσως. Θα έλεγα ότι η συνάντηση σήμερα θα μας επιτρέψει να μελετήσουμε τα πράγματα από κοινού και να μπορέσουμε αποτελεσματικά να καταλήξουμε σε συστάσεις που θα επιτρέψουν στις γυναίκες της Μεσογείου να φτάσουν σε μια ανάπτυξη και εξέλιξη προσωπική και επαγγελματική που θα τους επιτρέψει να συμβάλλουν περισσότερο στην ανάπτυξη των χωρών τους και να καταπολεμήσουν τη φτώχεια, την άγνοια, όλες τις πηγές συγκρούσεων στον κόσμο. Θα θέλαμε το καθεστώς ε, του Μαρόκου σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορέσει να συγκεκριμένει λίγο για να ανοίξουν νέες προοπτικές ανάπτυξης για να εξασφαλιστεί μια ε, κοινωνικο-οικονομική ε, εξέλιξη σίγουρη με την γυναική συμμετοχή. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Thank uh, Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Βανταρού. Στο τέλος της συνεδρίασης, αν δεν υπάρχουν τόσες πολλές ερωτήσεις και έχουμε πρόσθετο χρόνο, θα σας ζητήσω να αναπτύξετε περισσότερο τα σημεία της παρουσίασής σας. Τώρα η δεύτερη ομιλήτρια, Νεντέρα Σαμλού, που εκπροσωπεί την Παγκόσμια Τράπεζα ως ανώτερη σύμβουλος ε, Chief Economist για τη Μέση Ανατολή και την περιοχή της Βόρειας Αφρικής. Κυρία Σαμλό, έχετε τον λόγο. Και έχετε μια παρουσίαση νομίζω με θέματα, με διαφάνειες. Ε, έχετε τον λόγο. Well, good afternoon and... Ε, Καλό σας απόγευμα και ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση και διοργάνωση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτής της πολύ σημαντικής εκδήλωσης αυτής της συνεδρίας... ώστε να τεθεί στην ημερήσια διάταξη το θέμα των γυναικών σε αυτή την πολύ σημαντική συγκυρία. Αυτό που θα ήθελα να σας παρουσιάσω σήμερα είναι μια πολύ, ένα πολύ μικρό τμήμα μιας μελέτης ε, που αυτή τη στιγμή στην Παγκόσμια Τράπεζα ε, εκπονούμε και να σας δείξω κάποια αριθμητικά στοιχεία. Αν δεν γνωρίζουμε αυτά τα αριθμητικά στοιχεία δεν γνωρίζουμε το μέγεθος του προβλήματος ή το μέγεθος της λύσης σε αυτά τα προβλήματα. Θα ήθελα επίσης ίσως ε, να επιστήσω την προσοχή σε σχέση με την αισιοδοξία που κάποιοι μπορούν να έχουν γύρω από το γεγονός ότι πιστεύουν πολλοί ότι πρόκειται για μια νέα εποχή που διανοίγεται για τις γυναίκες στη Μέση Ανατολή. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να εισαγάγω κάποια από τα στοιχεία τα οποία ίσως ήδη έχετε δει και γνωρίζετε. Θέλω να ζητήσω πρώτα συγγνώμη για τα πολύ μικρά γράμματα στην εκτύπωση όπως παρουσιάζονται στις διαφάνειες. Αυτά που βλέπετε σε αυτή την πλευρά τώρα αυτών των στοιχείων είναι η τεράστια αύξηση όσον αφορά την παιδεία και εκπαίδευση των γυναικών πού βρισκόντουσαν οι γυναίκες το 1980 και πού βρίσκονται το 2000. Σε 20 χρόνια ο ταχύτερος, ο ταχύτερος ρυθμός ανάπτυξης ε, των, ε, της παιδείας των γυναικών, της εκπαίδευση των γυναικών σε σχέση με άλλες περιοχές. Ακόμα και σε άλλες ε, περιοχές υπήρξε άκρηση, αλλά όταν φτάνουμε στην συμμετοχή στον χώρο εργασίας μόνο 20-26% σημειώθηκε το αριθμητικό μέγεθος. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και συγγνώμη αν ομιλώ με μεταχείριση ρυθμό και θέλω να διασφαλίσω ότι θα μπορέσουμε να φτάσουμε ως το τέλος αυτής της παρουσίασης έγκαιρα. Αν δει κανείς το ποσοστό χρήσης ε, του ανθρώπινου δυναμικού των γυναικών βλέπουμε ότι στη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική αυτό το μέγεθος ε, είναι αυτή η γραμμή όπου θα έπρεπε να βρίσκονται και Βρισκόμαστε κάτω από τη γραμμή αυτή σχεδόν παντού και υπολογίζεται το δυναμικό με βάση το μέσο όρο όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό για τα, τα κέρδη όσον αφορά την ε, εκπαίδευση και παιδεία, την μείωση της ε, γονιμότητας ε, και όσον αφορά και τη δομή του πληθυσμού. Σε νέο πληθυσμό περισσότερες γυναίκες θα έπρεπε να συμμετέχουν στον, στην ηλικιακή αυτή, στο ηλικιακό φάσμα, ενώ αντίστροφα αν είναι πιο ο πληθυσμός, ε, μικρότερο το ποσοστό. Αυτό σε σχέση με τη Μέση Ανατολή και σε σχέση με τις άλλες ε, χώρες που βρίσκονται κάτω από, αυτό, από τον μέσο όρο. Πολύ λίγα άλλαξαν μεταξύ 1980 και 2001. Αυτό που θα ήθελα να σας παρουσιάσω υπό τους όρους ε, της, των πρόσφατων τεκμηρίων είναι μια διερεύνηση νοικοκυριών σε σχέση με τη Μέση Ανατολή θέλαμε να δούμε σε σχέση με το ΑΕΠ και τους δείκτες αυτούς ώστε να δούμε ε, σε σχέση με τα στοιχεία αυτά που είναι συγκρίσιμα όσον αφορά τις διάφορες χώρες και γίνονται πιο σύνθετα όσον αφορά περιοχές ε, ε, κάποιας χώρας όπου υπάρχει πιο κοσμοπολιτικός και σύνθετος χαρακτήρας. Επιλέξαμε μεταξύ Κάιρου και Σανά ώστε να έχουμε μια προσέγγιση σε σχέση με τη Μέση Ανατολή. Μια μεγάλη χώρα, μια μικρή χώρα, μια μεσαία χώρα, μια πλούσια, μια φτωχή είχαμε μεταξύ πολλών ανδρών και γυναικών δειγματοληπτικά της, ε, την έρευνα αυτή. Βλέπουμε ότι συνολικά ε, αυτό το οποίο βρήκαμε και ένας από τους κύριους στόχους ήταν να βρούμε ποιοι είναι οι πιο σημαντικοί λόγοι που έχουν επίπτωση στις γυναίκες στη συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας. Και εδώ είναι τα στοιχεία που θα ήθελα να συνοψίσουμε ε, μεγάλο αριθμό στοιχείων σε σχέση με τα όσα εμείς ε, ε, διερευνήσαμε. Αυτό που βρήκαμε είναι ότι σε μεγάλο βαθμό σε αυτές τις τρεις πόλεις, ναι, σε σχέση με την παιδεία, την εκπαίδευση των γυναικών, είναι σημαντική αλλά σε πολύ ψηλό επίπεδο, όταν είναι υψηλού επίπεδου. Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση δεν θα δώσει στις γυναίκες τη δυνατότητα να απασχοληθούν στην αγορά εργασίας. Και αν δει κανεί σε σχέση με τις χώρες αυτές, θα δει κανεί σε σχέση με το Αμάν, το Κάιρο και την Σανά ότι οι γυναίκες ακόμα και με υψηλότερη εκπαίδευση μπορούν να έχουν παντρευτεί και να μην εργάζονται. Αυτό που βρήκαμε είδαν ότι ουσιαστικά μόνο το υψηλότατο και πολύ υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης είναι εκείνο που έχει επίπτωση και οδηγεί τις γυναίκες στο να απασχοληθούν. Το αντίστροφο εκείνο, το αντίθετο εκείνο που είδαμε και μας ανησυχεί είναι ότι ο θεσμός του γάμου πραγματικά είναι ένα πολύ σημαντικό κόλλημα για να εργαστούν οι γυναίκες. Όχι τα παιδιά. Ναι, τα παιδιά κάπως είναι και αυτά ένα σφραγμός, ένα εμπόδιο. Αλλά το σημαντικότερο είναι ο γάμος. Και αυτό επειδή έχουμε τα θέματα της μητρότητας, την διάρκεια της γονεϊκής άδεια όσον αφορά την άδεια μητρότητας. Αλλά πρέπει να το δούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά τα θέματα τα οποία συνδέονται με το θεσμό του γάμου τη διαπραγματευτική ισχύ που έχει αυτό το ε, στοιχείο, αυτός ο συντελεστής και το τι δημιουργεί ως επιπτώσεις. Θα ήθελα να πω δύο λόγια παραπάνω για αυτό το θέμα των προδιαγραφών, των διατάξεων όσον αφορά το θεσμό του γάμου και ποιες επιπτώσεις ε, έχει. Όταν δούμε τη συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό των γυναικών, μια ερώτηση ε, διατυπώσαμε σε σχέση θα συμφωνούσατε με τις γυναίκες εκτός ε, του νοικοκυριού και την παρουσία τους ε, στον δημόσιο χώρο. Οι γυναίκες, ακόμα οι άνδρες και οι γυναίκες θα συμφωνούσαν με τέτοιου είδους εργασία και βρήκαμε ότι σε νοικοκυριά όπου δεν υπήρχε αντίρρηση ουσιαστικά αφορούσε αυτό τη συμμετοχή των γυναικών στο, ε, στην εργασία. Σε σχέση με τον οικοκυριό υπήρχε κάποια αντίρρηση. Όταν κάποιος ε, από τον οικοκυριό έλεγε ότι δεν μου αρέσει η συμμετοχή των γυναικών στην, ε, στο εργατικό δυναμικό, η επιλογή των οικονομικών ευκαιριών οδηγούν σε ένα πολύ μεγάλο φάσμα θα έλεγα. Θα ρώταγε κανείς γιατί, ποιος είναι εκείνος ο οποίος έχει αντιρρήσεις και ποιος ε, έχει ενστάσεις. Πρώτα απ' όλα το επίπεδο ενστάσεων ή αντίρρησης είναι το επίπεδο αντιρρήσεων των ανδρών στο αμάν το επίπεδο των αντιδράσεων και της άρνησης των γυναικών στο αμάν μετά των ανδρών στο Κάιρο η διαφορά του μπλε και του κόκκινου είναι η απάντηση ναι, μπορούν να εργαστούν οι γυναίκε υπό συγκεκριμένου όρου και προποθέσει Το μπλε. Το κόκκινο όχι. Δεν μπορούν να εργαστούν υπό, κανένα, υπό καμιά προπόθεση. Είδαμε στο Κάιρο το επίπεδο άρνηση ε, των γυναικών στο να συμμετάσχουν στο, σε εργασίε από του άνδρες ήταν πάρα πολύ υψηλό. Αντιδρούν οι άνδρες ε, και δεν θέλουν να εργάζονται οι γυναίκες εκτό νοικοκυριού. Η, θέση, η στάση των γυναικών βελτιώθηκε σημαντικά, αλλά στο Κάιρο είναι ενδιαφέρον να δει κανεί ακόμα και την άρνηση τη αντιρρήση των γυναικών να εργάζονται οι γυναίκες εκτός του νοικοκυριού τους, εκτός τη οικογένειάς τους. Ο πιο σημαντικός ρόλος και λυπούμε που σας βομβαρδίζω με όλες αυτές τις λεπτομέρειες ουσιαστικά είναι το ότι πρόκειται για αρχές ε, δεν εργάζεται η γυναίκα εκτός ε, νοικοκυριού. Εδώ έχουμε και το θέμα της ε, σεξουαλικής όχλησης, το ότι δηλαδή η, ε, ε, εξισορροπεί τα πράγματα η οικογένεια και δεν πρέπει η γυναίκα να ε, βγαίνει εκτός οικογένειας και δεν υπάρχει και η ανάγκη, δεν πρέπει να υπάρχει και η ανάγκη να εργάζεται εκτός οικογένειας διότι όταν, υπάρχουν, όταν βλέπουμε ότι το ποσοστό των οικογενειών εκείνων που έχει αρκετό εισόδημα είναι όμως μικρό αυτό είναι ενδιαφέρον να δει κανείς το θέμα της ε, αντιμετώπισης σεξουαλικής ε, όχλησης. Ε, γυναίκες δεν εργάζονται εκτός οικογένειας λοιπόν. Είναι πάρα πολύ συντηρητική αυτή η τοποθέτηση. Οι γυναίκες ανησυχούν για το πώς θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν όλα αυτά τα προβλήματα. Αυτή οι δύο, τα άλλα δύο στοιχεία, λυπούμε που σας δίνω τόσες πολλές λεπτομέρειες, είναι η αντίρρηση ανδρών και γυναικών όσον αφορά εισοδήματα, διαστρωμάτωση εισοδηματικών τάξεων και κατηγοριών. Αυτό που θα ήθελα να σας δείξω είναι η αντίρρηση νεότερων ανδρών. Ηλικιακή ομάδα, εδώ έχουμε τους άνδρες και εδώ έχουμε τις γυναίκες. Και η αντίρρηση των ανδρών, των νεότερων ανδρών ηλικιακά, οι ίδιοι αυτοί οι νέοι άνδρες που πιστεύουμε και θεωρούμε ότι είναι έχουν πρόσβαση στα, στην κοινωνία της πληροφορίας και των ηλεκτρονικών έχουν αντιρρήσει στο να εργάζονται οι γυναίκες εκτός οικογένειας. Και αυτό είναι ανησυχητικό. Δύο τρίτα του πληθυσμού στη Μέση Ανατολή και στην Αίγυπτο είναι κάτω από ε, τα 30 χρόνια ηλικιακά. Οι άνδρες λοιπόν είναι αυτοί που έχουν αντιρρήσεις. Οι νέοι είναι πολύ πιο συντηρητικοί από ότι οι γονείς τους και είναι πολύ πιο συντηρητικοί στην τοποθέτησή τους. Να μην είναι αναμένουμε κάποια θαύματα αν μέσω μιας δημοκρατικής διαδικασίας δούμε να υπάρχουν συντηρητικά ρεύματα ή συντηρητικές ε, θέσεις και τάσεις. Αυτοί είναι ε, οι ε, νέοι εκείνοι οι οποίοι θα έχουν ακριβώς αυτό το πιο συντηρητικό ας το πούμε έτσι πλαίσιο αντίδρασης από ότι οι γονείς τους και η αντίρρηση σε σχέση με τις γυναίκες στο να εργάζονται είναι ακριβώς περίπου θα έλεγα αν, μέχρι και το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και στο ε, πανεπιστημιακό επίπεδο. 20% από το δειγματοληπτικό αυτό ε, ποσοστό έχουν την ε, πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Εκείνοι λοιπόν που θα πήγαιναν και να ψηφίσουν για το Σύνταγμα είναι εκείνοι οι οποίοι θα βρίσκονται σε αυτό το πεδίο εκπαίδευσης. Και αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι είναι πάρα πολύ συντηρητική πάρα πολύ συντηρητική. Θα ήθελα να σας το αναφέρω αυτό. Υπάρχει το ερώτημα και ρωτάνε κάποιοι, ίσως κάποιοι από αυτούς που έχουν αντιρρήσει στο να εργάζονται οι γυναίκες είναι εκείνοι που είναι άνεργοι. Βλέπουμε ότι εκείνοι που είναι κατά το, του να εργάζονται οι, οι γυναίκες 50% στο ΑΜΑΝ, 65% στο Καϊρό, 54% από αυτούς έχουν εργασία, ε, δεν είναι άνεργοι. Αυτή είναι η δομή που προτιμούν να έχουν μεγαλύτερη επιρροή όσον αφορά την οικογένεια ως άντρες. Δεν είναι οι αντιρρήσεις που να προέρχονται σε σχέση με κάποιους ανέργους αυτό το οποίο θα ήθελα να σας δώσω ως μήνυμα και δεν θέλω να περάσω σε λεπτομέρειες σε όλα τα συμπεράσματα είναι το θέμα του αν οι γυναίκες θα υποφεληθούν πραγματικά από αυτή την ε, ε, εξουσιοδότηση που θα οδηγήσει τις γυναίκες να συμμετάσχουν, να αλλάξει ο ρόλος των γυναικών στο τέλος τέλος. Τώρα βλέπουμε όμως ότι όταν θα έχουμε το θέμα των ψηφοφοριών και της ε, έγκρισης ε, ε, πολιτικών κομμάτων ή συντάγματος θα πρέπει να δούμε τι είναι εκείνο που η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Παγκόσμια Τράπεζα μπορεί να πράξει και να συνεισφέρει από πλευράς της ώστε να αποφύγουμε αυτή την εξέλιξη πραγμάτων. Δηλαδή να μην έχουμε κάτι το οποίο θα αποβεί εις βάρος των γυναικών στο τέλος τέλος. Ευχαριστώ. Thank uh, uh, Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και αν κάποιος από την Παγκόσμια Τράπεζα δεν, θα, δεν ερχόταν να μας ε, δώσει κάποια τέτοια στοιχεία, εμείς θα είμαστε οι πρώτοι που θα παραπονούμαστε. Και σας ευχαριστούμε για αυτό που κάνατε. η κυρία Μπαντάου θα πρέπει να έχει πέντε λεπτά μετά την επόμενη παρουσίαση για κάποιες διευκρινήσεις. Είναι δύσκολο να είναι πάντα ο πρώτος που παρεμβαίνει ως αγορητής και σίγουρα περισσότερα πράγματα θέλουμε να μάθουμε από εσά. Επιπρόσθετα θέλω να σας υπενθυμίσω υπέρ της διαφάνειας και του ανοιχτού χαρακτήρα αυτού αυτής της ε, εκδήλωσης όλα τα σεμινάρια, workshops ε, βρίσκονται στο δικτυακό τόπο και όλα θα είναι διαθέσιμα ε, ηλεκτρονικά από το διαδίκτυο και από το website. Και αν χρειάζεστε κάποιες λεπτομέρειες μπορώ να σας τις δώσω περαιτέρω λεπτομέρειες κατά το τέλος της συνεδρίασης. Τώρα έχω ιδιαίτερη χαρά να καλέσω την τρίτη που θα παρέμβει από πλευράς μας και είναι η κυρία Κακάινεν που είναι ε, υπάλληλο στο Ευρωπαϊκό Κέντρο κατάρτιση. Θα παρουσιάσει τι δραστηριότητε αυτής, τη της ε, υπηρεσίας Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την πρόσβαση των γυναικών στην εκπαίδευση, στην κατάρτιση, στην ε, εκπαίδευση. Έχετε τον λόγο παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν είναι μόνο η Παγκόσμια Τράπεζα που μπορεί να σας δώσει στοιχεία εγώ δεν γνώριζα τα σχετικά με την δική σας παρουσίαση και ίσως μπορεί να υπάρχει και κάποια επικάλυψη σε σχέση με τις δύο μας παρουσιάσεις. Ελπίζω επίσης όμως ότι θα αλληλοσυμπληρώνονται οι παρουσιάσεις μας, οι παρεμβάσεις μας εκπροσωπώ το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Κατάρτισης, ε, ένα ε, νέο θεσμό που ε, δραστηριοποιείται όσον αφορά την εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα παρουσιάσω τα αποτελέσματα μελέτης που έχει γίνει σε σχέση με την κατάρτιση και εκπαίδευση, σε σχέση με τις γυναίκες και την απασχόληση για, αυτές για αυτή την περιοχή και για αυτές τις χώρες. Εμείς επικεντρωθήκαμε ιδιαίτερα σε νεότερες γυναίκες, σε νέες γυναίκες γυναίκες από τα 15 έως τα 29 έτη ηλικιακά. Επίσης ε, είχαμε και εξετάσαμε ε, όσον αφορά τον ιδιωτικό τομέα το, τη συνιστόσα των ε, εργοδοτών. Για να παρουσιάσω το πλαίσιο αυτής της τοποθέτησης και παρουσίασης ως θέμα σε αυτό το σεμινάριο, η εκπαίδευση και η παιδεία διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο όσον αφορά την επανάσταση στην Αραβική Άνοιξη είναι εκείνο που ε, δίνει την δυνατότητα στο να μπορούν να διαβάζουν, ε, να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, σε πληροφορίες ε, αυτοί, αυτές οι γυναίκες, να είναι σε θέση να διαδραματίσουν ρόλο διεκδικώντας τα δικαιώματά τους, να διαδραματίσουν ένα ρόλο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για τη δημοκρατία και όπως και σε σχέση με την προηγούμενη παρουσίαση θα ήθελα να πω ότι είναι η χρονική συγκυρία για αλλαγή, αλλά δεν θα πρέπει να είμαστε υπερβολικά αισιόδοξοι. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε σχέση με τις, την πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά την εκπαίδευση και την κατάρτιση των γυναικών σε αυτή την περιοχή και να μπορέσει να αντανακλάται στη συμμετοχή των γυναικών, στο εργατικό δυναμικό και στην απασχόληση, που είναι ένας τρόπος να δώσουμε δικαιώματα στις γυναίκες. Δεν θεωρούμε ότι όλες οι γυναίκες ή όλοι οι άνδρες πρέπει να εργάζονται υποχρεωτικά, αλλά αν αποφασίσουν να εργαστούν θα πρέπει να έχουν ίσα δικαιώματα και ίδια δικαιώματα να έχουν αξιοπρεπή απασχόληση και εργασία όπως και οι άνδρες. Έτσι λοιπόν δεν θα επαναλάβω αυτά τα οποία αναφέρονται στο αυξημένο επίπεδο εκπαίδευσης ε, κατάρτισης ε, στο πρωτογενές και ή δευτεροβάθμιο ε, επίπεδο για γυναίκες και άντρες. Απλά και μόνο να αναφέρω ότι στην τριτογενή, τριτοβάθμια εκπαίδευση μπορούμε να δούμε μια εξέλιξη σημαντική έναντι της Ευρώπης. Είναι εκπροσωπούνται περισσότερο οι γυναίκες σε σχέση με τους άντρες. Αυτό αναφέρθηκε και από άλλους που παρενέβησαν σήμερα το απόγευμα ως στοιχείο, για παράδειγμα σε σχέση με την Ευρώπη. Ωστόσο, όπως προαναφέρθηκε σε αυτή την περιοχή, το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναμικό είναι από τα χαμηλότερα σε παγκόσμια κλίμακα. Αν κάνουμε σύγκριση με άλλες περιφέρειες και περιοχές όπου σημειώθηκε μείωση ε, και έχουν, ε, υπάρχει μια τάση όσον αφορά τη συμμετοχή των γυναικών στο εργασιακό δυναμικό και κάποιες, και, κάποιες εξελίξεις δικτών όμως ε, δεν ήταν δυνατόν στην νότια όχθη της Μεσογείου να υπάρξει κάποια ριζοσπαστική αλλαγή. Η συμμετοχή στο εργασιακό δυναμικό ανάλογα με την εκπαίδευση, το επίπεδο εκπαίδευσης αυξάνεται και ιδιαίτερα το υψηλό επίπεδο ε, εκπαίδευσης, ε, η τριτοβάθμια εκπαίδευση δίνει πραγματικά αυτό το δυναμικό. Οι άνδρες συμμετέχουν στο εργασιακό δυναμικό άσχετα όμως από το επίπεδο ε, εκπαίδευσης ή μόρφωσης ή εξειδίκευσης τους. Παρ' όλα αυτά σε αυτή την περιοχή βρισκόμαστε όπου η ανεργία των νέων είναι πάρα πολύ υψηλή και αυτό έχει συνεισφέρει και αυτό ως στοιχείο στην ε, Αραβική Επανάσταση που ξεκίνησε και από αυτούς τους άνεργους και τη δυσαρέσκεια. Πρέπει να δούμε όμως ε, γιατί και ενώ τα ποσοστά ανεργίας και των γυναικών και των ανδρών αυξάνονται το επίπεδο ανεργίας των γυναικών είναι πάντα ανώτερο από το επίπεδο ανεργίας των ανδρών ποσοστία. Και σε σχέση και με τα στοιχεία που έχουμε από το ε, Ίδρυμα Κατάρτισης ε, σε σχέση με την Παγκόσμια Τράπεζα, εδώ έχουμε δύο μεγέθη. Πρώτον για την Νότια και Ανατολική Μεσόγειο. Η μία συνιστώσα αντανακλά το, ποσοστό, το ενεργό ποσοστό στο ποσοστό απασχόλησης ή απασχολησιμότητας ανδρών και γυναικών. Και το άλλο από κάτω είναι ο μέσος όρος των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ βλέπει κανείς ένα συγκρίσιμο στοιχείο. Το θέμα της συμμετοχής των γυναικών και της απασχόλησης τους, απασχολησιμότητάς τους, αρχίζει από ένα χαμηλότερο ποσοστό εκπαίδευσης. Ωστόσο υπάρχει μια διαφορά. Ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει μια παρόμοια τάση σε σχέση με άνδρες και γυναίκες ότι δηλαδή το ποσοστό συμμετοχής ε, όταν αναζητούν ή ψάχνουν να βρουν μια ε, θέση εργασίας οι άνδρες και οι γυναίκες αυξάνονται οι πιθανότητες με την εκπαίδευση και το ίδιο συμβαίνει με την απασχολησιμότητα. Στην Νότια και Ανατολική Μεσόγειο βρισκόμαστε σε χαμηλό επίπεδο. Το βλέπετε αυτό, αυτό αντανακλά το υψηλό ποσοστό εκπαίδευσης ε, των γυναικών σε σχέση με τη συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας. Υπάρχει όμως αυξανόμενο χάσμα, αυξανόμενο κενό μεταξύ της κόκκινης ε, και της ε, ελαφρά μπλε γραμμής όσον αφορά την ανεργία των γυναικών που αυξάνει περισσότερο σε σχέση και με την εκπαίδευσή τους. Άσχετα σε σχέση με τις, τα προσόντα ή τα διπλώματα και πτυχία. Είναι η αρνητική διακριτική μεταχείριση συλλήβδιν που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες όσον αφορά την αγορά εργασίας. Τι θα έπρεπε εδώ, πώς θα έπρεπε να αντιδράσουμε σε αυτό έχουμε χαμηλή, ε, χαμηλή επιστροφή όσον αφορά τις ε, επενδύσεις ε, στην οικονομική ζωή όσον αφορά την εκπαίδευση. Βλέπουμε δεν εκμεταλλεύονται το ανθρώπινο δυναμικό σωστά. Δεν είναι δυνατόν να το εκμεταλλευτούμε σωστά. Έχουμε υψηλό ποσοστό εξάρτησης από έναν εργαζόμενο οικογένεια. Οι γυναίκες δεν συμμετέχουν, βρίσκονται πολύ χωλένουν οι γυναίκες όσον αφορά την συμμετοχή τους στην ε, εργασιακή ζωή και έτσι υπονομεύεται η προσπάθεια καταπολέμησης της φτώχειας. Σύντομα θα ήθελα να αναφερθώ στα αποτελέσματα αυτής της, ε, του, του οργάνου μας. Είμαστε ένα όργανο σε σχέση με την έρευνα της ε, ε, κατάρτισης και τα θέματα αγοράς-εργασίας εργαζόμαστε και στην Κεντρική Ασία, υποψήφιες προς ένταξη χώρες και στη Νότια και στην Ανατολική Μεσόγειο γενικότερα οι γυναίκες και οι δυνατότητες, οι προοπτικές απασχόλησης. Στόχος είναι να προαχθεί η ισότητα των ευκαιριών όσον αφορά την εργασία μεταξύ ανδρών και γυναικών τριετές πρόγραμμα το επίκεντρο είναι ε, σε ιδιωτικό τομέα ε, λόγω των, ε, της επικέντρωσής μας σε αυτές τις χώρες επίσημη ε, τυπική αγορά εργασίας και όχι άτυπη αγορά εργασίας που δεν παρέχει τα ίδια δικαιώματα ούτε παρέχει προσφέρει συνταξιοδοτικά δικαιώματα ή γονεϊκή άδεια και γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε ότι η επίσημη οικονομία είναι εκείνη η οποία μπορεί να παράσει στις γυναίκες αξιοπρεπή απασχόληση και στις τρεις ε, περιπτώσεις ε, ε, Αίγυπτο, Ιορδανία και την Ισία, όπως είπα, το επίκεντρο ήταν η εξέταση της μεταβατικής περίοδου από το σχολείο στην επαγγελματική απασχόληση νέων γυναικών από 15 29 ετών. Και έχουμε και δειγματοληπτική έρευνα όσον αφορά και την συνιστόσα των εργοδοτών, ιδιαίτερα όσον αφορά τις νέες γυναίκες και βλέπουμε ότι έχουμε και τον τομέα των, ε, της υπαίθρου. Κύριος στόχος μας ήταν στο να δούμε ποιο είναι το δυναμικό αυτών των τομέων για να απασχοληθούν οι γυναίκες και αν δεν απασχολούνται γυναίκες ε, να δούμε ποιο είναι το πρόβλημα, αν υπάρχει πρόβλημα προσφοράς και ζήτησης και τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να δημιουργηθεί ένα πιο εποφελές πλαίσιο από πλευράς της ε, κατάρτισης και εκπαίδευσης για τις γυναίκες κάποια συμπεράσματα, πολύ σύντομα θα αναφέρω κάποια. Αυτό που είδαμε στον τομέα του τουρισμού, οι γυναίκες ε, λιγότερο εκπροσωπούν όσον αφορά τον μέσο όρο εκπροσώπησης ε, των γυναικών σε άλλους τομείς ε, απασχόλησης βλέπουμε ότι σε πόλεις βρισκόντουσαν πιο υψηλά στην εκπροσώπησή τους ε, οι γυναίκες. Αυτό που είδαμε είναι ότι στις εταιρείε ICT υπήρχε μια θετική τάση, μια θετική εξέλιξη ένα έτος πριν από την ε, ε, έρευνα αυτή είχαν ποσοστία απασχολήσει περισσότερες ε, γυναίκες ε, οι επιχειρήσεις αυτές. Στον τουρισμό ήταν το αντίθετο το οποίο διαπιστώθηκε. Λιγότερες γυναίκες προσελήφθησαν από, σε σχέση με τις ICT εταιρείες. Υπάρχει όμως εδώ και η εξή παρατήρηση. Είναι ένα τομέα που δεν προσελκύει μόνο γυναίκε από το υψηλότερο ε, μερίδιο εκπαιδευμένων και κατατισμένων γυναικών που είπαμε ότι έχουν τη μεγαλύτερη συμμετοχή, η, πιο, ε, η υψηλότερη εκπαίδευση γυναίκε. Βλέπουμε όμω ότι υπάρχει και η τάση να απασχολούνται εκεί σε αυτόν τον τομέα γυναίκε με χαμηλότερα προσόντα. Οι γυναίκε υποπροσωπούνται λοιπόν και αν δει, λοιπόν την, κανείς την ε, προσφορά όσον αφορά τις γυναίκες, οι γυναίκες ε, σε σχέση με τις ε, δραστηριότητες ICT που βλέπουμε ότι είναι πανεπιστημιακού επίπεδου. Όμως λιγότερες γυναίκες υποβάλλουν τις, καταθέτουν αιτήσει να προσληφθούν σε αυτόν τον τομέα. Υπάρχει έλλειψη γυναικών όσον αφορά την ε, προθυμία τους να απασχοληθούν, να σε αυτόν τον τομέα, ιδιαίτερα του τουρισμού, λόγω του ότι υπάρχει αρνητική, αρνητικός προειδεασμός όσον αφορά το να εργάζεται η γυναίκα σε κάποια συγκεκριμένα επαγγέλματα, τα οποία δεν θεωρούνται ιδιαίτερα τιμητικά εντός εισαγωγικών για αυτές, ιδιαίτερα σε κάποιες περιοχές ε, της χώρας. Όσον αφορά την πρόσληψη, η μεταβατική αυτή περίοδος σε σχέση με τις προσωπικές επαφές και συστάσεις που είχαν ακόμα έχουν πολύ μεγάλο ρόλο αυτές οι επαφές και συστάσεις. Ε, συνδέονται λιγότερο με κοινωνικά δίκτυα οι γυναίκες επειδή έχουν πολύ πιο περιορισμένο εύρος επαφών και δραστηριοτήτων είναι περιορισμένες στον νοικοκυριό τους και δεν έχουν δυνατότητες άλλων επαφών. Τώρα εξειδικεύοντας το φύλλο όσον αφορά την ε, απασχόληση βλέπουμε ότι υπάρχουν προκαθορισμένα ας το πω έτσι ε, πλαίσια ενώ αυτό δεν είναι νόμιμο και βλέπουμε ότι υπάρχουν συγκεκριμένα επαγγέλματα στα οποία διαπιστώνεται αυτή η τάση. Στο επίπεδο λοιπόν δραστηριοποίησης επαγγελματικά των γυναικών επικεντρώνονται περισσότερο στο marketing, στην διοίκηση, στο software οι γυναίκες και πολύ λιγότερο σε ε, ε, ηγετικές θέσεις. Γυναίκες σε σχέση με το ε, hardware λένε ότι ενώ μπορεί να έχουν τα προσόντα όσον αφορά τα, το hardware, οι εργοδότες προτιμούν να απασχολούν τις γυναίκες σε θέσεις ε, software. Τώρα, προκλήσεις ε, όσον αφορά το συνδυασμό επαγγελματικής ζωής ε, και οικογενειακής ζωής. Μη σεβασμός και μη συμμόρφωση με την εργασιακή νομοθεσία Πολλές ε, φορές ε, είναι αυτό ένα θέμα το οποίο δημιουργεί προβλήματα. Όμως, καμιά φορά αποφεύγεται με το να μην απασχολούν περισσότερο από 300 για παράδειγμα γυναίκες διότι εκεί αυτό είναι το δεδομένο ε, όριο το οποίο πρέπει να τους αναγκάζει να σέβονται συγκεκριμένα δικαιώματα. Μετά το θέμα των δυνατήτων εκπαίδευσης για μια απασχόληση. Οι εργοδότες ξέρουν ότι οι γυναίκες φεύγουν από την θέση εργασίας τους όταν ε, επενδευτούν και γι' αυτό δεν προτίθενται να επενδύσουν τόσο πολύ σε εκπαίδευση ε, στην, ε, στον τόπο εργασίας. Μετά, η αρνητική κοινωνική ιδέα, όχι μόνο από την κοινωνία γενικά, αλλά από τα μέλη της οικογένειας. Τους ε, αδελφούς, τους πατέρες ε, και οι γυναίκες που αναζητούν επίσης μοντέλα να ακολουθήσουν, ε, δεν έχουν πολλούς που να έχουν πετύχει μια τέτοια θέση και να μπορούν να τους δεσμεύσουν. Μετά, το θέμα της μεταφοράς, ε, των χωρών εργασίας, σεξουαλική ε, παρενόχληση, προκλήσεις για τις εταιρείε τώρα που αποσχολούν τις γυναίκες, το οικονομικό κόστος. Ε, δεν είναι όλα αυτά αρκετά για να προστατευτούν οι γυναίκες στην νομοθεσία αν οι ιδιωτικέ επιχειρήσεις είναι μόνε που αντιμετωπίζουν το κόστος απασχολή γυναικών. Υπάρχουν επίσης οργανωτικά προβλήματα, γιατί πρέπει να υπάρχουν διαφορετικέ καφετήριε, διαφορετικά μέσα μεταφορά. Επίσης το θέμα ότι οι εργοδότες θεωρούν ότι το να απασχολούν γυναίκες ε, δίνουν μια καλύτερη εικόνα της επιχείρησης αλλά όχι όσον αφορά το θέμα της επαφής με τους πελάτες. Τι μπορεί να γίνει λοιπόν. Θα δώσω κάποιες συστάσεις, έχω ένα λεπτό στη διάθεσή μου ακόμα, τι μπορεί να γίνει, ιδίως στον τομέα της εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης. Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες βέβαια. Η πρόθεση της εικόνας της γυναίκης που εργάζεται από τα ΜΜΕ και αλλιού να υπάρχει ε, κατεύθυνση επαγγελματική που να λαμβάνει υπόψη το φύλλο και να δίνονται οι σχετικές πληροφορίες των δυνατοτήτων της απασχόλησης και ενθάρρυνσης των γυναικών να αναλάβουν μη παραδοσιακές γυναικείες ε, θέσεις απασχόλησης και να ενθαρρυνθούν οι άντρες από την άλλη μεριά να αναλάβουν θέσεις παραδοσιακά γυναικείες ούτως ώστε το καθώς αυτών των θέσεων να υψωθεί. Επίσης να αποθαρρυνθεί ε, η δημιουργία στερεοτύπων στα σχολεία που έχουν επιδράσει στην κοινωνία, η πρακτική κατάρτιση των γυναικών, να υπάρχουν δυνατότητες κατάρτιση των γυναικών που σπουδάζουν, παραδείγματος χάρουν, και ιδίω σε περιβάλλον ε, όπου συνεργάζονται άνδρες και γυναίκες και η υποστήριξη των γυναικών να ενσωματωθούν στον τόπο της απασχόλησης και να μην υπάρχει έτσι διακριτική αρνητική μεταχείριση και σεξουαλική παρενόχληση. Η συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους. Παρακαλώ, μην βιάζεστε υπερβολικά, γιατί καλύτερο είναι να ακούσουμε τι έχει να μας πείτε παρά να έχουμε περισσότερες ερωτήσει. Συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους. Ε, θα ήταν καλό περισσότερες γυναίκες να συνεργάζονται στα συνδικάτα. Περισσότερα συνδικάτα σήμερα λαμβάνουν υπόψη τα δικαιώματα των γυναικών και προασπίζουν την εργασιακή νομοθεσία που υπάρχουν για τον σεβασμό και των εργασιακών δικαιωμάτων των γυναικών. Δεν είναι δηλαδή σημαντικό μόνο η κυβέρνηση να συνεργαστεί με τους ιδιωτικούς εργοδότες, αλλά και τα συνδικάτα. Και θα πρέπει τα συνδικάτα να προωθήσουν περισσότερους, περισσότερες δυνατότητες στις πρόσφυξης των δικαιωμάτων των γυναικών. Όπως είπα προηγουμένως, δεν θα πρέπει μόνο ο ιδιωτικός τομέας να έχει το βάρος της απασχόλησης των γυναικών. Για να ξεπεραστεί αυτό θα ήταν δυνατό πούμε, να δοθούν φορολογικά κίνητρα στις ιδιωτικές επιχειρήσεις να απασχολούν περισσότερες γυναίκες και να συμμερίζονται το κόστος της φροντίδας των παιδιών, της μεταφοράς και της άδειας Δεν θέλω να ε, χρονοτριβούσε ιδιαίτερα. Ένα λεπτό λέει ο πρόεδρος. Εντάξει, ένα λεπτό. Ίσως στην αρχή ήμουν κάπως αρνητική, αλλά τελευταία ε, έχω να σας πω ότι υπάρχει μια ελπίδα που βλέπω εγώ σήμερα. όταν πήγαμε στην Εθνισία για να κάνουμε τη μελέτη επιτόπου το 2008, αναζητώντας πληροφορία, στατιστικά στοιχεία, πήγαμε στην την Ένωση Δημοκρατικών Γυναικών που εκπροσωπούνται σήμερα. Αλλά αυτό που έγινε συνεδρία ήταν ότι ψιθυρίζαμε. Γιατί ακριβώς η Ένωση αυτή φοβόταν μήπως ε, κάποιος κατέγραφε αυτές τις συζητήσεις. Και είμαι πάρα πολύ ευτυχή σήμερα που είδα ότι μπορούμε να μιλήσουμε ανοιχτά μεγαλόφωνα, με μικρόφωνα και να συζητούμε όλα τα πράγματα ανοιχτά. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Um, Ευχαριστώ για την παρουσίασή σας, όπως είπα. Θα δώσω άλλα πέντε λεπτά στην κυρία Μπαντράουι για να συμπληρώσει αν θέλει κάτι σε αυτά τα οποία ακούσαμε. Έχουμε μαζί μας τώρα την αξιότιμη Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την κυρία Κράτσα. Σας καλωσορίζουμε εδώ. Λοιπόν, κυρία Μπαντράουι, έχετε το λόγο. Λοιπόν, σε σχέση με αυτά που είπε η κυρία εδώ δίπλα μου, που ανησυχούσε λίγο για το ποσοστό συμμετοχής της γυναίκας στην οικονομική ανάπτυξη της ε, περιοχής. Με τις μεταρρυθμίσεις που βλέπουμε σήμερα, με τις δημοκρατικές αλλαγές, μπορούμε να δείξουμε ότι υπάρχει πράγματι ένας κάποιος δισταγμός και μια παράδοση η οποία βαραίνει θα έλεγα τις κοινωνίες του νότιου τμήματος της Μεσογείου. Στην παρουσίασή μου εγώ αναφέρθηκα στην αρχή των ποσοστώσεων και θα ήθελα να επανέλθω στην αρχή αυτή λέγοντας ότι είναι πράγματι ένα μέσο το οποίο μπορεί να βοηθήσει να αλλάξουν οι νοοτροπίες η ποσόστοση. Η Αιγυπτία φίλη που ήταν εδώ πριν είπε ότι θα ήταν προτιμότερο η γυναίκα μόνη της να αρπάξει τα δικαιώματα που της ανήκουν. Αλλά παρόλα αυτά ε, θα πρέπει να ζούμε σε μια κοινωνία ανοιχτή που δέχεται τις αλλαγές. Αλλά όταν μιλάμε για μια κοινωνία παραδοσιακή που δεν θέλει να αλλάξει τον τρόπο ζωής της και που θέλει να κρατήσει τη γυναίκα στο σπίτι, τότε η ποσόστοση μπορεί να είναι ένα μέσο το οποίο θα βοηθήσει την γυναίκα να καταλάβει τη θέση της στα κοινοβούλια και στα διοικητικά συμβούλια. Εγώ είμαι υπέρ, υπέρ λοιπόν των ποσοστώσεων, το είπα και στην παρουσίασή μου η ποσόστοση ίσως είναι μια ενδιάμεση λεγόμενη περίοδος για να αλλάξουν οι νοοτροπίες, να επικρατήσουν τα δικαιώματα της γυναίκας. Μια απλή παρέμβαση λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε λίγα λεφτά για το τελευταίο θέμα που θέσατε. θα ήθελα να πω ότι σε σχέση με το θέμα γενικότερα της ισότητας, τα ποσοστά απασχολησιμότητας των γυναικών αλλά και των μειονοτήτων, μία από τις πιο προοδευτικές χώρες στην Αφρική είναι η Ρουάντα. Είναι γνωστό ότι έχει το υψηλότερο ποσοστό γυναικών στο κοινοβούλιο και στην πολιτική γενικότερα. Έχουμε λοιπόν ένα καλό παράδειγμα εδώ και όλα όσα συζητήσαμε σήμερα το απόγευμα οι περισσότερες από τις χώρες μας χρειάστηκε να τα αντιμετωπίσουν. Υπάρχουν λοιπόν μέθοδοι για να ξεπεράσουμε τα προβλήματα τα οποία έχουμε, να υπάρξει πολιτική βούληση, να εντοπίσουμε το πρόβλημα και να το λύσουμε. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω σήμερα το απόγευμα όλες σας για τις εξαιρετικές παρεμβάσεις τις οποίες κάνατε, για το θάρρος το οποίο επιδείξατε και την προσπάθειά σας γενικότερα. Αυτό με διαβεβαιεί ότι βρισκόμαστε στον σωστό δρόμο και θα πετύχουμε τον στόχο μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Now, uh, uh, Λοιπόν, αυτά υπάρχει κάποιο πολύ σύντομο σχόλιο, ερώτηση, οποιοδήποτε είναι εδώ, αλλά σύντομα. Πάντα χρειάζεται ένας πρώτο πόρος, δεν ξέρω ποιος έχει το θάρρος να κάνει μια ερώτηση ή ποια. Καλώς λοιπόν, αυτό δείχνει ότι όλες οι ερωτήσεις σας έχουν ήδη απαντηθεί. Είμαστε σίγουροι για τον τρόπο που θα εξελιχθούν τα πράγματα. Θα ήθελα να πω στους οργανητές αυτές της συνάντησης. Α, έχετε το λόγο φυσικά. Μία ερώτηση στις ε, δύο γειτόνισές μου. Παρουσίασαν και οι δύο κάποιες μελέτες, μία της Παγκόσμιας Τράπεζας και μία από το ETF που είχαμε πολύ χαρά να συνεργαστούμε μαζί τους, το Μαρόκο ποτέ δεν θεωρήθηκε χώρα στόχος για αυτές τις μελέτες. Πάντα σε αυτές τις μελέτες εκπροσωπούνται οι ίδιες συνεχώς χώρες και θα ήθελα να σας προσκαλέσω να προχωρήσετε και σε στατιστικές μελέτες και στη δική μου χώρα. Πράγματι πολύ καλή εξαιρετική παρατήρηση και θα ζητήσω από τη συνάδελφο από την Παγκόσμια Τράπεζα, δεν ξέρω αν θέλει να απαντήσει, αλλά παρόλα αυτά ε, είμαι παρόν στην πρόσκληση που απευθύνεται, δεν ξέρω αν θέλουν να πούν κάτι οι συνάδελφοι. Ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Είναι καλό να ξέρουμε ότι είστε εκεί όταν σας χρειαζόμαστε. Προσπαθήσαμε να ελέγξουμε τη μεθοδολογία της μελέτης αυτής. Βρισκόμαστε σε μια πρώτη φάση ελέγχου των υποθέσεων. Το Μαρόκο έχει πολλές ομοιότητες αλλά και πάρα πολλές διαφορές. Η δομή, ο πολιτισμός ε, είναι εντελώς διαφορετικά από τις υπόλοιπες χώρες και θα πρέπει να περιμένουμε και διαφορετικά αποτελέσματα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση πάντως η κυρία Καϊκίνεν. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Με μεγάλη χαρά θα ανταποκριθούμε να διευκρινίσω ότι όταν κάνουμε τέτοιες μελέτες το κάνουμε μετά από, τη, από αίτημα των χωρών εταίρων αν θέλετε. Δεν επιβάλλουμε εμείς μελέτες στις διάφορες χώρες Η επόμενη προγραμματική περίοδος για την μελέτη μας έχει σαν βασικό στόχο την ισότητα των φύλων. Και γι' αυτό θα ζητήσουμε πληροφορίες και από σας. Ευχαριστώ. Πριν περάσουμε στην κυρία Αντιπρόεδρο για να κλείσει την συνάντηση, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όσους οργανώσατε τη συνάντηση αυτή. Εμείς δεν αγγίξαμε παρά την επιφάνεια του προβλήματος. Υπάρχει μια περιπλοκότητα και πολυπλοκότητα των καταστάσεων τις οποίες αντιμετωπίζουν οι γυναίκες. Ακριβώς επειδή είσαστε γυναίκες υφίσταστε προβλήματα, διακρίσεις. Σκεφτείτε να ήσασταν επίσης ε, γυναίκα ανάπηρη και να υφίσταστε διακρίσεις λόγω των θρησκευτικών σας πεπιθήσεων ή λόγω του γενετήσιου σας προσανατολισμού. Υπάρχουν πάρα πολλά επίπεδα εν πάση περιπτώσει καταπίεσης και πρέπει να απευθύνουμε την πολιτική μας αποφασιστικότητα σε όλες τις ε, περιπτώσεις που χρειάζεται γιατί αν δεν το κάνουμε έστω και σε μία περίπτωση ακυρώνουμε την προσπάθεια που κάνουμε σε όλες τις άλλες περιπτώσεις. Λοιπόν, θα δώσω στην Αντιπρόεδρό μου ε, τον λόγο η οποία προσωποποιεί την αποφασιστικότητα επιτυχίας των στόχων που όλοι επιδιώκουμε. Η κυρία Κράτσα Τσαγκαροπούλου έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, Κύριε Πρόεδρε αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί εταίροι της Νοτιοόχθης της Μεσογείου, με ενθουσιασμό και συγκίνηση έρχομαι μεταξύ σας εδώ στο εργαστήριο αυτό εργασίας λόγω της ουσιαστικής σημασίας του θέματος της συμμετοχή των γυναικών. Είναι ουσιαστική στην πρόοδο αυτής της ε, περιοχής ε, που βρίσκεται σε μετάβαση στην ε, Μεσόγειο και στην Μέση Ανατολή όπου υπάρχει έντονος άνεμος βούλησης για ένα καλύτερο μέλλον και προσωπική και συλλογική συμμετοχή για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός. Καταρχήν επιτρέψτε μου να σας ευχαριστήσω όλους και όλες για τη συμμετοχή σας στο εργαστήριο αυτοεργασίας. Ιδίω εσά, εσάς κύριε Πρόεδρε για τον ενθουσιασμό με τον οποίο συνοδεύσατε αυτή την πρωτοβουλία είναι τιμή για το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο να μπορεί να δεχθεί στις, ε, στο κτίριό του γυναίκες από Σόγιο δυναμικές και δεσμευμένες σε μία καρποφόρο ανταλλαγή ιδεών και απόψεων. Οι, οι εικόνες των γυναικών από την Αίγυπτο, την Λιβύη, τη Συρία που διαμαρτύρονται για να πετύχουν καλύτερη μοίρα όπως τις είδαμε στις ε, πλατείες τους, στους δρόμους τους ανά τον κόσμο, μας οδήγησαν σε πολύ συγκίνηση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αμέσως υποστήριξε αυτή τη βούληση μεταρρύθμισης και τοποθετήθηκε στο πλευρό των πληθυσμών που δεσμεύτηκαν στην άγουσα της ανανόησης της δημοκρατικής. Αυτό που μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση στην επανάσταση του Ιωσενιού, όπως παραδείγματο χάρη στην ε, Αίγυπτο την ημέρα του θύμου είναι ότι τα στερεόπιτη παπουσίων για τους άνδρες, τις γυναίκες, τις μειονότητες τέθηκαν κατά μέρο ούτω ώστε να υπάρχει μια κοινή πρόσκληση προς την δημοκρατία, προς το σεβασμό των βασικών δικαιωμάτων και ένα μέλλον με ελπίδα και αξιοπρέπεια μίας και καθενός. Τα πρόσφατα γεγονότα καταδεικνύουν λοιπόν ξεκάθαρα ότι η φωνή της τολμηρής και γραφερής γυναίκας δεν μπορεί να παραβλεφθεί. Για πολύ καιρό οι γυναίκες ήταν θύματα της έλλειψης της ε, ελευθερίας σε αυτές τις χώρες της Μεσογείου και της Μεσοανατολής και ήταν περιορισμένος όσον αφορά τα λόγια τους και τη δυνατότητα εξέλιξής τους στις κοινωνίες αυτές θα πρέπει τώρα να γίνουν πλήρες συμμετέχουσες στην συνοχή, την ειρήνη και την ανάπτυξη των χωρών τους. Επιτρέψε μου να τονίσω εδώ την υποστήριξη και την αλληλεγγύη που θα πρέπει να δείξουμε σήμερα προς τις γυναίκες της Λιβύης και της Συρίας των οποίων η μάχη είναι ιδιαίτερα ηρωική τα δικαιώματα της γυναίκας, όπως και γενικά ο σεβασμός των βασικών δικαιωμάτων, αποτελούν εκ των όνους ουκ άνευ και είναι απαραίτητες για τη δημοκρατία και την ποιότητα ζωής. Είναι σημαντικό να συνεχίσουμε προς την ίδια άγουσα και να συγκεκρινοποιήσουμε τις προσπάθειές μας, ούτως ώστε να αρθούν τα ε, εμπόδια που υπάρχουν στα πολιτιστικά νομικά, πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά συστήματα για να εξασφαλιστεί η συμμετοχή της γυναίκας στην αγορά εργασίας σε όλους τους επαγγελματικούς τομείς και σε όλα τα επίπεδα λήψη αποφάσεων. Αυτά τα προβλήματα με ενδιαφέρουν όλους ιδιαίτερως και από αυτή την οπτική ε, γωνία είχα ήδη τη δυνατότητα το 2002 να παρουσιάσω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια έκθεση σχετικά με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι των χωρών της Μεσοφίου όσον αφορά την προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών και την ισότητα των ευκαιρών στις λόγους χώρες. Αυτός ο στόχος της ισοτομίας είναι το κλειδί της πλήρους συμμετοχής και συμπερίληψης των γυναικών στην διαδικασία πρόθεση πολιτικής σε όλα τα επίπεδα και όσον αφορά την τοπική πολιτική και όσον αφορά την δημόσια δίδυξη, όσον αφορά το κοινοβούλιο, όσον αφορά την κυβέρνηση και όσον αφορά και τις διεθνείς οργανώσεις και τις οργανώσεις της ε, κοινωνίας των πολιτών. Οι νέες γυναίκες που είχαν τη δυνατότητα να εκφραστούν μέσω των κοινωνικών μέσων και να παρουσιάσουν τις απόψεις τους θα μπορέσουν να προωθήσουν ακόμα περισσότερο αυτά τα μέσα. Βλέπουμε ένα δυνομισμό που, που συνοδεύει την εξέλιξη των παραδοσιακών ΜΜΕ διευκολύνοντας τη μεταφορά στη δημοκρατία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρώτος δωρητής ε, βοήθεια στις ε, χώρες της Μεσογείου. Θέλει να υποστηρίξει τη δημιουργία συγχρόνων κοινωνιών δημοκρατικών που σέβονται τις βασικές αρχές. Τα μέσα της βοήθειας της ε, ε επικοδομικής της ενίσχυσης είναι πολλές. Επενδύσεις σε όλους τους τομείς καταρχήν. Παραδείγματος χάρη επίσης με το πρόγραμμα Ευρωμέτ Audiovisual η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει τον οπτικοστοκουστικό και κινηματογραφικό τομέα των χωρών εταίρων. Αυτοί οι δύο τομείς αποτελούν έναν ε, ε, δημιουργικό τομέα ανάπτυξης και μια σημαντική πηγή εκπαίδευσης. Προωθούμε επίση την κοινωνικο-οικονομική εξέλιξη και μια πληροριστική εξέλιξη στην περιοχή αυτή αν κάτι τέτοιο χρειάζεται για την δημοκρατική μετάβαση. Για να εγγυηθούμε την αποτελεσματικότητα των ΜΜΕ υπάρχει μια στενή συνεργασία μεταξύ των ε, εργαζομένων στο τομέα αυτό και από τις δύο χθέσεις της Μεσογείου. Η πρόθεση της ιδέας της ειρήνης και της ε, ε, συμμετοχής στην Μεσόγειο μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την ουσιαστική ενίσχυση των ΜΜΕ. Έτσι, εγώ, ως αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που είμαι υπεύθυνη για την ενημέρωση και την εκπαίδευση και επίσης υπεύθυνη για τις σχέσεις Ευρωμεσογείου, Ευρω θα ήθελα να οργανώσω ένα σεμινάριο ευρωμεσογειακό για τους δημοσιογράφους με στόχο να προσεγγίσουν οι επαγγελματίες του τομέα των δύο οχθών της Μεσογείου για να δούνε ποια είναι τα προβλήματα και να ανακαλύψουν ποια είναι τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους για να μπορέσουν να ενημερώνουν πλήρως και ποιοτικά όλους τους πολίτες και όλους τους πολιτικούς της ε, ευρωμεσογειακής περιοχής για τις προκλήσεις που έχουμε αμοιβαία και τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να δράσουμε. Πράγματι, προετοιμάζεται μια σχετική πρωτοβουλία για να ενθαρρυνθεί, ενθαρρυνθεί η ελεύθερη έκφραση και να δημιουργηθεί ένας δημόσιος χώρος στο οποίο θα υπάρχει η απαραίτητη ανταλλαγή πληροφοριών και όπου θα δίνεται μια συνέχεια στην πολιτική και των δύο οχθών της Μεσογείου. Θα ήθελα όμως να τονίσω ότι μου φαίνεται ότι πάρα πολύ σωστό οι ίδιες οι γυναίκες να δράξουν τις ευκαιρίες που τους δίνουν τα πρόσφατα γεγονότα και η ευρωμεσογειακή συνεργασία ούτως ώστε να αναλάβουν τον νέο τους ρόλο, να προωθήσουν τα κεκτημένα δικαιώματα για να πετύχουν φιλόδοξους στόχους για την μοίρα τους, τη χώρα τους, την περιοχή τους. Που σήμερα βρίσκεται ενώπιον αποτελεσματικό ε, σημαντικών ε, στοιχείων για την ιστορία τους. Θα πρέπει να προωθήσουμε την ευημερία και την ε, ενσωμάτωση γειτονικών χωρών να δοθεί μια απάντηση στην κλίση για αλλαγή της πολιτικής όπου οι πολιτικές οι πολίτες συγγνώμη, θα βρεθούν πάνω από τις προκλήσεις και τις ε, Η διεθνή κοινότητα συμπεριλαμβανομένη τη Ευρωπαϊκή Ένωση υποστήριζε πάντα τη συμμετοχή των γυναικών στι αραβικέ χώρε και θα συνεχίσει να προωθεί αυτή την τόσο ουσιαστική τυχή της πολιτικής τους. Θα πρέπει από τη συνάντησή μας εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή των ε, Δικαιωμάτων Γυναικών και την Επιτροπή ε, των ε, Εξωτερικών Υποθέσεων είχαμε μία συνάντηση με την κυρία Μπασλέ που είναι τώρα διευθύντρια στο Ηνωμένα Εθνή υπεύθυνη για την ισότητα των φύλων μέσα στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών. Στις 24 Μαρτίου είχαμε τη συνάντηση αυτή και συμφωνήσαμε για μια συνεργασία που θα επιτρέψει χεραφέτηση των γυναικών και υπέρβαση των στερεοτύπων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και είναι ξεπερασμένα αλλά ευρεωμένα στις αραβικές κοινωνίες και μια ανανέωση της ισότητας ανδρών και γυναικών. Έτσι, το κοινοβούλιο μας ε, δέχθηκε πολύ θετικά την απόφαση για την εξασφάλιση των στόχων της Επανάστασης έχοντας κατά νου την εγκαθίδρυση ενός ισομερού συστήματος για τις επόμενες νομοθετικές εκλογές στην νησία. Ελπίζω ότι και οι άλλες χώρες περιοχής εκείνης, ακόμα και οι ευρωπαϊκές χώρες, θα ακολουθήσουν αυτό το πολύ τολμηρό παράδειγμα που πολλά υπόσχεται για τη μακροπρόθεσμη εξέλιξη και που θα αυξήσει έτσι συμμετοχή των γυναικών στα μελλοντικά πολιτικά συστήματα. Τέλος, είναι υποχρεωσή μας να εξασφαλίσουμε η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι εργασίες των ιδρυμάτων, πολιτικών κομμάτων, συνδικάτων και μη κυβερνητικών οργανώσεων που εργάζονται πάνω στις σχέσεις με τις χώρες της Μεσογείου και της Μεσοανατολής να τονίσουν το πόσο επίγουσα είναι η εγκαθίδρυση μιας κοινωνίας χωρίς διακρίσεις που βασίζεται στο φύλλο ή κατά άλλων μειονοτήτων. Τέλος, θα πρέπει να υπάρχουν επίσης μέτρα που θα υποβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ισομερής συνέλευση για την Μεσόγειο και η Επιτροπή της για τα Δικαιώματα των ε, Γυναικών θα πρέπει να ασκήσει τις ε, υποχρεώσεις για να μπορέσει να επιτευχθεί ο στόχος αυτός. Συμμετέχουμε με ενθουσιασμό στις εργασίες αυτής της ε, Επιτροπής, της Ισομερούς, της Ισομερούς Συνέλευσης, όπου συνεργάζονται οι βουλευτές από τα ε, εθνικά κοινοβούλια ε, χωρών και από τις δύο όχθες της Μεσογείου. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, ακρόασαν αυτοί που είχαμε σήμερα, που με μεγάλη ευχαρίστηση υποδεχθήκαμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι σημαντικές σε αυτή την ιστορική στιγμή. Μας επιτρέπουν να συναντηθούμε, να ανταλλάξουμε απόψεις, να συζητήσουμε επικοδομητικά με στόχο να δημιουργήσουμε μία κοινωνική κοινή ε, συνείδηση και να δώσουμε στις γυναίκες τον, τη θέση που τους αρμόζει σε όλες τις σύγχρονες κοινωνίες και μέσα στο πλαίσιο όλων των σχεδίων των κοινωνιών μας. Σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας, για τη συμβολή σας στην τόσο επικοδοματική και σας υπέσχομαι να επαναλάβω αυτό το ραντεβού. Ευχαριστώ. Thank you, Σας ευχαριστούμε κυρία Πρόεδρε. Ήταν εξαιρετικά αυτά τα συμπερασματικά τα οποία μας εκφράσατε και έτσι εμπνευσμένοι θα περάσουμε στην βραδιά αυτή. Θέλω να ευχαριστήσω για το ε, σεμινάριο αυτό όλες σας και θέλω να ευχαριστήσω για το εξαιρετικό του έργο και τους διερμηνείς. Ολοκληρώσαμε τις εργασίες μας. Καλό σας βράδυ.